Καλώ och eh, ήλθατε. Θα συνεχίσω στα σουηδικά. Όποιο δεν καταλαβαίνει σουηδικά, ίσω πρέπει να βάλει τα ακουστικά του. Ελπίζω λοιπόν ότι περάσατε ένα καλό μεσημέρι, είχατε μια καλή μεσημεριανή διακοπή και είχατε επαρκή όρεξη, γιατί περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της διάσκεψής μας. Το πρώτο τμήμα της απογευματινής συνεδρίασης αφορά το θέμα και α, μόλις, μόλις επανήρθε η κυρία Πιέτη Κάινερ γιατί ένιωθα κάποια ανησυχία είναι το θέμα γυναίκες στην πολιτική, προώθηση της ισότητας των φύλων για τους πολιτικούς στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις και το δεύτερο τμήμα του απογεύματος θα αφορά το θέμα της προώθησης της ισότητας των φύλων στην νομοθεσία και θα είναι παρούσα μεταξύ μας η κυρία Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Πιέτη Κάινεν. Υπάρχουν κάποιοι που είχαν ζητήσει από το πρωί να λάβουν το λόγο και για αυτού που θέλουν το απόγευμα επίση να λάβουν το λόγο θα ακολουθήσουμε την ίδια ακριβώ διαδικασία όπως το πρωί. Με μεγάλη χαρά λοιπόν χαιρετίζω την κυρία Πιετικάινεν. Υπήρξατε εισηγήτρια για μια εξαιρετικά κατά την άποψή μου σημαντική έκθεση η οποία κρίση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία και η οποία αφορά το θέμα της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικούς ε, φορείς και κοινοβούλια και κυβερνήσει. Και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και την θερμή σας συνεργασία κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια που είχα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης εκθεσής μου ήταν εξαιρετικά σημαντική και μου δώσανε πολύ σημαντικά σχόλια και συνεισφορές για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Να ξεκινήσω με τον τίτλο, με την επικεφαλίδα της εκθέσεως. Οι γυναίκες στην πολιτική, τα θέματα ισότητος και ανισότητος, στην εκπροσώπηση. Οι γυναίκες δεν έχει χειρότερες λήπτριες αποφάσεων από τους άνδρες, αλλά ούτε και το αντίθετο. Ούτε οι άνδρες, ούτε οι γυναίκες είναι καλύτεροι, έχουν το προνόμιο της καλύτερης γνώσης ή κρίσης. Δεν νομίζει κανείς ότι η ικανότητα ξεκινάει από τα χρωμοσώματα και από το φύλλο στο οποίο ανήκει ο καθένας και ούτε θεωρεί κανείς ότι η εμπειρία που αποκτούν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους είναι λιγότερο σημαντική από αυτή που αποκτούν οι άνδρες. Το θέμα λοιπόν της ισιότητος σημαίνει ότι θέλουμε και οι γυναίκες που αποτελούν το ίμιση του πληθυσμού να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων. Θέλουμε την εμπειρία ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσματος γυναικών στη στάθμιση και λήψη αποφάσεων. Η ισότητα επίσης σημαίνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανθρώπινα δικαιώματα. Το ξαναλέω, τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί στις συζητήσεις μας πολλές φορές τίθεται το ερώτημα του κατά πόσο τα θέματα ισότητας των γυναικών πρέπει να την χάνουν των ίδιων νομοθετικών διασφαλίσεων όπως άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Και φαίνεται σαφές σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις λόγω φυλής, λόγω θρησκείας, σεξουαλικών προτιμήσεων ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλου λόγου. Αλλά για κάποιο λόγο στις συζητήσεις μας εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενο το, πώς, το κατά πόσο τα δικαιώματα των γυναικών βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα δικαιώματα των ανδρών και με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα τώρα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών στην Ευρώπη. Αυτό διαφαίνεται και από τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν πρόκειται να επανέλθω γιατί σας έχουν δώσει τα στοιχεία ήδη από το πρωί και καταλαβαίνετε πόσο υπολείπονται γυναίκες εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν τούτου, όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο το οποίο ατενίζεται, τόσο μικρότερη είναι η εκπροσώπηση των γυναικών όταν βλέπετε προεδρίες επιτροπών, όταν βλέπετε υπουργικού θόκους κτλ. Όλο και λιγότερες είναι γυναίκες. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα αριθμητικό θέμα μονάχα, ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το θέμα της, ε, της διακρίσεως των διαφόρων μορφών εξουσίας. Είναι η μακρά σκιά της πατρικής και της μητρικής εξουσίας. Οι άντρες θέλουν να έχουν τον έλεγχο πάνω στους υλικού πόρους. Είναι άνδρες πρωθυπουργοί, άνδρες υπουργοί οικονομικών, άνδρες υπουργοί βιομηχανίας. Πολλές φορές οι γυναίκες πρέπει να περιορίζονται σε μορφές εξουσίας που ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται κάποιοι πόροι, παραδείγματος χάρη παιδεία, υγειονομική περίθαλψη, περιβάλλον. Αυτό από μόνο του, ο διαχωρισμός θέσεων εξουσίας, δημιουργεί ήδη μία ανισότητα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τρία ζητήματα. Πρώτον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα το αριθμητικό. Πόσε γυναίκε βρίσκονται στην πολιτική. Δεύτερον, πρέπει να δούμε σε τι είδου θέσει έχουν ευθύνη οι γυναίκες. Και το τελευταίο θέμα είναι το θέμα του αυτόφωτου ή όχι των γυναικών. Το θέμα του ηλίου και της σελήνης. Αν μπορούν οι γυναίκες από μόνες τους να λάμπουν χωρίς να αντανακλούν φως από κάποιον άλλο. Έχουμε στην Επιτροπή Γυναικών ένα πρόεδρο που είναι άνδρας και τρεις γυναίκες που είναι αντιπρόεδροι. Αλλά πάντα οι γυναίκες είναι αντιπρόεδροι, αντισυντονιστές, ε, υπό εισηγητές. Κάτι, έχουν πάντα μια δευτερεύουσα θέση. Όταν βλέπουμε λοιπόν το θέμα της ισότητας, δεν πρέπει να το δούμε μοναχα ποσοτικά πρέπει να κοιτάξουμε πιο ενδελεχώς και ποιοτικά. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τις θέσεις οι οποίες είναι πραγματικά ηγετικέ, όπως η θέση ενός Πρόεδρου, από τις αναπληρωματικά ηγετικέ θέσεις, όπως είναι η θέση του χάρη μιας Αντιπροέδρου. Θα έρθω μετά στις προτάσεις μας για το τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση είναι γεγονό ότι πρέπει να έχουμε μια πιο συστηματική και πολυεδρική αντιμετώπιση για όλα αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν επιρροή για τα θέματα αυτά. Οι αντιλήψει καταρχήν, ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνδρες και οι γυναίκε, πώ παρουσιάζονται από τα μέσα ενημέρωση οι άνδρες και οι γυναίκες όταν δρουν στην πολιτική, ποιε είναι οι οικονομικέ και κοινωνικέ δυνατότητε που ανοίγονται για του άνδρες και τι γυναίκε και πόσο ίσε είναι ποιες είναι οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ενεργειών τους, πώς δουλεύουν οι κομματικές δομές, πώς δουλεύουν οι νομοθετικές δομές για να επιτρέψουν και να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών ή όχι. Ένα βασικό λοιπόν πλέγμα θεμάτων που είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να προχωρήσουν περισσότερο είναι τα θέματα του πώς λειτουργεί μια κοινωνία και κατά πόσο διευκολύνει την λειτουργία στην πολιτική. Όσο πιο θετικά είναι αυτά τα πλαίσια, τόσο πιο πολύ διευκολύνουν, τόσο περισσότερο διευκολύνουν την παρουσία των γυναικών σε θέσεις εξουσίας. Σε ό,τι αφορά την αμοιβέ, είναι πολλές φορές το 70% μονάχα η αμοιβή των γυναικών από ότι εναντί των ανδρών. Και στο βιομηχανικό τομέα οι γυναίκε εργάζονται συνήθω σε γυναικείε σε εισαγωγικά εργασίε, οι οποίε είναι πιο κακοπληρωμένε από τι ανδρικέ. Τίνουν ακόμα οι γυναίκε να έχουν το μερίδιο του λέοντος σε ό,τι αφορά την παιδική φροντίδα και την οικογενειακή φροντίδα. Οι γυναίκες μένουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι και περισσότερα χρόνια πολλές φορές στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι οι καριέρες τους υποφέρουν και οι αποδοχές τους υπολείπονται των ανδρικών αποδοχών. Σε οικονομικό επίπεδο λοιπόν είναι σε υποδέστερη θέση και είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτές να ασχοληθούν με την πολιτική και να έχουν έναν ενεργό ρόλο σε σχέση με τους άντρες. Αν δούμε επίσης το πλήρες φάσμα ηλικίας στη ζωή μιας γυναίκας, οι γυναίκες έχουν χαμηλότερες συντάξεις γιατί η καριέρα τους έχει προχωρήσει πολύ λιγότερο και έχουν μείνει πιο πολύ χρόνο στο, σπίτι τους, επομένως οι συντάξεις τους είναι πολύ μικρότερες από αυτές των ανδρών. Επομένως, ένα προαπαιτούμενο για την ισότητα θα πρέπει να είναι η ισότητα αποδοχών. Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σύστημα πρόνοιας στην κοινωνία. Και γι' αυτό έχω ρίξει το σύνθημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει ο καλύτερος φίλος των κοριτσιών. Αν είχαμε υπηρεσίες που θα έδιναν φροντίδα για τους ηλικιωμένους, βρεφονιπιακούς σταθμούς και όλα αυτά, αυτό θα ελάφραν τις γυναίκες από την ανάγκη που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκλειστικό, αποκλειστική υποχρέωση των γυναικών να φροντίζουν τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουμε να συζητούμε περισσότερο για την κοινωνική διάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλει στους πολίτες της η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους άνδρες και στις γυναίκες που είναι πολίτες της, το δικαίωμα να έχουν ένα βασικό ελάχιστο εισόδημα όταν δεν έχουν άλλη πηγή ε, προσόδων και ορισμένες βασικές υπηρεσίες. Φυσικά αυτό αντιμετωπίζεται διαφορετικά από κάθε κράτος μέλος και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάλογα με την φάση της ζωής που βρίσκεται ο καθένας σε σχέση με το τι είναι το απαραίτητο ελάχιστο εισόδημα ή οι απαραίτητες ελάχιστες ε, υπηρεσίες αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει εγγεγραμμένο στο Σύνταγμα κάθε χώρας το δικαίωμα σε κάποιο ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών και κάποιο ελάχιστο εισόδημα εάν δεν έχει κανείς άλλη πηγή εισόδηματος. Τώρα, σε σχέση με τις θέσεις ευθύνης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η ανισότητα σε σχέση με τις αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Εδώ αναφέρομαι στις λεγόμενες θετικές δράσεις. Ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι πρέπει να υπάρχει μια ανάλυση για, την, για τον αντίκτυπο στα δύο φύλλα σε οποιασδήποτε ενέργειες και να έχουμε μια σειρά δράσεων για να μπορούμε να αυξήσουμε την συμμετοχή των γυναικών σε επίπεδα ευθύνης. Εκλεγμένες θέσεις τώρα. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα, το ευρωπαϊκό επίπεδο, το δημοτικό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο. Στη συζήτησή μας ξεκινήσαμε με το θέμα των πολιτικών κομμάτων. Γιατί για μας το πρόβλημα, μάλλον ο πυρήνας της πολιτικής δράσης βρίσκεται στα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα σε όλα τα επίπεδα να εξασφαλίσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών, για να μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια μεγαλύτερη ισότητα σε επίπεδο αξιωμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα να έχουν στο καταστατικό τους και στους διαδικαστικούς κανόνες την αρχή της ισοτιμίας. Όταν υπάρχει λοιπόν η εκλογή των ε, υπευθύνων και των ηγετών θα πρέπει να υπάρχει ισότης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών. Αυτή η αρχή λοιπόν ότι τα καταστατικά και οι κανόνες διαδικασίες των κομμάτων είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι εθνικά θα πρέπει να έχουν αυτή την αρχή της ισοτιμίας, αυτό θα πρέπει να είναι και ένα προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε δημόσια χρηματοδότηση κομμάτων σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο. Ένα δεύτερο θέμα αφορά τις εκλογές. και έχουμε συζητήσει για το θέμα προτιμησιακών συστημάτων στις εκλογές. Αυτό είναι δύσκολο να εναρμονιστεί γιατί έχουμε διαφορετικά συστήματα εκλογικά στις χώρες μας. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει την εναλλαγή ανδρών και γυναικών σε θέσεις ε, ε, πολιτικής ευθύνης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο εξασφαλίζει ότι υπάρχει ισότης σε ό,τι αφορά όχι μόνο τις θέσεις, αλλά και τα αξιώματα και τη δημοσιότητα που δίνεται σε άνδρες και γυναίκες. Αυτό από μόνο το όμως δεν φτάνει. Πρέπει να έχουμε και εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες. Επειδή οι γυναίκες αυτή τη στιγμή αμείβονται λιγότερο και είναι πολύ πιο δύσκολο για μια γυναίκα να βρει χρηματοδότηση για μια προεκλογική εκστατεία και επειδή έχει λιγότερη ορατότητα, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε θετική διάκριση, σε θετική δράση αυτή τη στιγμή. Πρέπει ένα τμήμα από τους πόρους που αποδίδονται για εκλογικές εκστρατείες να δίδεται μισιακά στις γυναίκες υποψηφίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σαρώσουν την πολιτική και να διώξουν τους άνδρες από την πολιτική, απλώς να μπορέσουμε να επαναφέρουμε μια ισορροπία να σταματήσει αυτή η κατάσταση που οι άνδρες δίνουν όλες τις πρωτοκλασσάτες εκλογικές μάχες και είναι στα μέσα ενημέρωσης και οι γυναίκες είναι σε δευτερεύον επίπεδο. Αυτό επίσης που κάναμε ήταν να στείλουμε επιστολές στα κόμματά μας και να τους ζητήσουμε να εξετάσουν το θέμα αυτό και να το φέρουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ μίλησα με τις ε, ε, γυναίκες συναδέλφους μου από τα φιλανδικά πολιτικά κόμματα, τους παρουσίασα τις προτάσεις μας και τους ρώτησα τι θα κάνουν για αυτό το θέμα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε όλοι στα κράτη-μέλη σας, να συλλέξετε τις απόψεις των συναδέλφων σας στα εθνικά κράτη και τις προθέσεις τους για να διορθωθεί αυτή η σημερινή κατάσταση. Ανεξάρτητα φυσικά από πολιτικές παρατάξεις. για τις εκλογές και τις επερχόμενες εκλογές. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία των φορέων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε πολύ καλές εμπειρίες για συνεργασία τέτοιων οργανώσεων, είτε είναι πολιτικού χαρακτήρα είτε όχι, που εργάζονται από κοινού σε πλατφόρμες. Για να θέσουν το θέμα της ε, ισότητας των φύλων εν ώψη των εκλογών και να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση των γυναικών για να υποστηρίξουν γυναίκες υποψηφίους. Οι εκστατείες αυτές ήταν αρκετά επιτυχής. Γιατί λοιπόν να μην διδαχτούμε από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουμε σε όλες τις χώρες μας πλατφόρμες αυτού του, ίδιου, του είδους από οργανώσεις γυναικών που μπορούν να συνεργάζονται με όλα τα πολιτικά κόμματα για να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση και να θέσουν τα θέματα ισότητος πριν από τις εκλογές και έτσι να υποστηρίξουν τις γυναίκες υποψηφίους. Να μπορεί λοιπόν να υπάρχει και μια εθνική χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε αυτές τις πλατφόρμες. Ελπίζω λοιπόν ότι και η Κομισιόν όταν προσεγγίζουμε τις επόμενες ευρωεκλογές και αυτό ετέθηκε στην πρωινή συζήτηση. Η Κομισιόν θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία θα χρηματοδοτεί την υποστήριξη της ε, ισότητας ευκαιριών και την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών στις εκλογές. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια σταθερή και συνεχιζόμενη εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υποστηρίζει πλατφόρμες γυναικείων οργανώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλοι μας ως εθνικοί βουλευτές, ως ευρωβουλευτές, ως υποψήφοι θα μπορούμε μέσω αυτών των πλατφορμών να ανταλλάσσουμε απόψεις. Μια πρόταση θα ήταν να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μια σύνδεση με το δικαστήριο της Χάγης και να εξεταστεί περισσότερο ο μηχανισμός με τον οποίο έχουν προωθηθεί οι θέσεις των γυναικών για τα θέματα αυτά. Και το δικαστήριο αυτό μπορεί να έχει στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και όταν μιλάμε για τα κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης, και εκεί πάλι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ε, συνεργασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δικτυακή πύλη μέσω της οποίας μπορούν οι γυναικείες οργανώσεις και οι πλατφόρμες να ανακαλύπτουν η μεν την δε και να μπορούν έτσι να συμμερίζονται ιδέες για δράσεις και εκστρατείες. Τώρα, φεύγουμε από τις εκλογές και πάμε τις ερετές ε, γυναίκες θέσεις ε, εκλεγμένες και τις ποσοστώσεις. Οι δικές μας ε, συστάσεις τι λέγουν από τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ήδη διαβουλευτεί και καταλήγουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος κανονισμού που να αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, που να ορίζει το εξής. Όταν πρόκειται για θέσεις διορισμένες ή εκλεγμένες, ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, πλήρης ισότητα στους αριθμούς για να σπάσει αυτή η διάκριση, ας πούμε, και στις οικονομικές επιτροπές, αλλά και σε επιτροπές ισότητας των φύλων. Θα πρέπει να έχουν ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Ε, ή και πρόεδρος, ας πούμε, εντός της επόμενης δεκαετίας ή δεκαπενταετίας. Όχι να είναι δηλαδή στις οικονομικές επιτροπές ε, πρόεδροι άνδρες και στις ε, επιτροπές ισότητας πρόεδροι γυναίκες. Επίση, θα πρέπει να υπάρχουν μέθοδοι και διαπραγμάτευσης που να εφαρμόζονται και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν εκλέγουμε αντιπροέδρους και προέδρους σε επιτροπές να υπάρχει ισότητα και, και στους αριθμούς. Αυτό το καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ένα κακό παράδειγμα ως προς την ίση εκπροσώπηση ε, σε ό,τι αφορά ε, το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι που βαραίνει τους ώμους της κυρίας Αγγελίλη αυτό το θέμα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά όχι τα αιρετά αξιώματα, αλλά τους διορισμούς. Είναι άλλη η μάχη που πρέπει να δώσουμε εδώ. Γιατί ε, στους διορισμούς και στα πόστα αυτά που ορίζονται ε, άνδρες ή γυναίκες, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι πρεσβείες, οι αντιπροσωπείες μας εκεί, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα υπόλοιπα αξιώματα ε, στη διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είτε είναι ε, υπουργεία σε εθνικό επίπεδο. Έχει σημασία να έχουμε εξασφαλισμένη την ίση προσώπηση. Γιατί ε, χρειάζεται ισορροπία στη λήψη των αποφάσεων και στο προκατακτικό στάδιο και στις προτάσεις που κατατίθενται για να λαμβάνουμε εμείς αποφάσεις. Και εκεί είναι ένα θέμα λοιπόν και ποιότητας και ισότητας. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν προτείνουμε να έχουμε αυτές ε, τις θετικέ δράσεις ε, και ε, στη δημόσια διοίκηση και στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. για να μπορούν οι γυναίκες να βοηθούνται στη σταδιοδρομία τους, δηλαδή να έχουν κατάρτιση και εκπαίδευση για διοίκηση, για ε, ε, ηγετικέ θέσει, ε, να μην υπάρχει αυτή η γυάλινη, η κρυστάλλινη οροφή όπω ονομάζεται, να σταματάει κάπου η ανέλυξη των γυναικών επειδή δεν έχουν τα προσόντα ή τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα για να γίνουν managers ή να αναλάβουν ηγετικά αξιώματα και ότι από ένα επίπεδο και μετά μόνο άνδρες μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Επίσης, στις προτάσεις μας Ε, συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προτείνουν δύο υποψηφίους για επίτροπο, έναν άντρα και μία γυναίκα. Γιατί εμείς ζητούμε να υπάρχει ισότητα στον αριθμό των ε, ε, επιτρόπων, αλλά τα κράτη-μέλη προτείνουν. Αν δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες, πώς να εξασφαλίζεται αυτό. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να προτείνουν έναν άντρα και μία γυναίκα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες θέσεις όπου τα κράτη-μέλη ορίζουν υποψηφίους. Και εκεί η σύστασή μας είναι η εξής. Ας πούμε, σε ένα ορίζοντα δεκαετίας θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ίση εκπροσώπηση, δηλαδή να ε, προτείνουν έναν υποψήφιο άντρα και μία γυναίκα για τις διάφορες θέσεις ε, και τα αξιώματα, τα ηγετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου διορίζονται οι ε, υποψήφοι. Γιατί και πάλι θα έχουμε τεράστιες διαφορές και στην εκπροσώπηση εδρών γυναικών. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, ε, μικρότερες ίσως, πολλές, αλλά για να έχουμε χρόνο και για συζήτηση, να σας αναφέρω τι κάνουμε αυτό το καιρό και τι σχεδιάζουμε. Ωραία. Έχουμε αυτή την έκθεση που διαπιστώνει αυτά που σας είπα και στείλαμε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του θέτουμε υπόψη αυτά που προτείνουμε Επίσης, επιστολή στείλαμε στον κύριο Φαν Ρόμποϊ. Ξέρετε ότι τα θέματα ισότητας ουδέποτε απασχόλησαν ε, την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε υψηλό επίπεδο και συζητούμε από τον κύριο Φαν Ρόμποϊ να συζητηθούν και αυτά. Ήδη απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βεβαίως επισήμως απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου έτσι κι αλλιώς και στα διάφορα πολιτικά κόμματα. Επίσης αποταθήκαμε, καθένα στα δικά του και στις πολιτικές μας ομάδες, για να ε, βεβαιωθούμε ότι στο μέλλον θα αλλάξουν οι κανονισμοί και τα καταστατικά των κομμάτων για να υπάρχει ίση ε, εκπροσώπηση και στις εσωτερικές ενδοκομματικές ε, εκλογές και των πολιτικών ομάδων όταν προτείνουν υποψηφίους για αξιώματα στο Κοινοβούλιο θα ήθελα να σας προτείνω μια εκστρατεία τώρα. Ε, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 50-50. Μισό-μισό. Από διάφορα πολιτικά κόμματα, λοιπόν, και το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ε, προέρχεται αυτή η πρωτοβουλία. Και τι σημαίνει. Αν έχουμε ε, αυτή την ομάδα σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο διακομματικά να προωθεί θέματα ισότητας να υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμός και ένα σημείο επαφής με την πλατφόρμα των γυναικείων οργανώσεων και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων και δράσεων διότι όλα αυτά είναι πιο αποτελεσματικά όταν γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στα διάφορα κράτη-μέλη ταυτόχρονα και έτσι μπορούμε ο καθένας να μαθαίνουμε από τον άλλον τι συμβαίνει στα διάφορα κοινοβούλια. Και τι κρύβεται εκεί ως ιδέα από πίσω ότι το θέμα θα είναι επόμενες ευρωεκλογέ και μπορούμε να αργήσουμε να κάνουμε αυτή την εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας πούμε να υπάρχει υποψήφιος ένας άνδρας και μια γυναίκα ε, αυτό θα ήταν από τα βασικά θέματα που θα κυριαρχούσαν, ας πούμε, για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Και θα ζητήσουμε από τους διάφορους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα στα κράτη-μέλη να το αναλάβουν και να το λάβουν υπόψη. Έτσι έχουμε και μια ευκαιρία να συναντιόμαστε, να αλληλοβοηθούμαστε σε διάφορες δραστηριότητε αυτής της εκστρατεία. Για παράδειγμα, να υπάρχει κάποια καθοδήγηση και υποστήριξη ε, γυναικείων υποψηφιωτήτων. Κυρίως για γυναίκες που πρωτοεμφανίζονται στην ευρωπαϊκή ε, σκηνή ας πούμε, και δεν ξέρουν πολύ καλά τα δημόσια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, υπομονή σας. Ε, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο περιεχόμενο όλο της έκθεσης και στις δράσεις, αλλά θεώρησα καλό για τη συζήτηση να μακρηγορήσω λίγο και να αναλύσω με περισσότερες λεπτομέρειες για να πάρετε έτσι μια γεύση των όσων κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Πιετικάινεν. Κατά την άποψή μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ανάλυση και η λεπτομερής παρουσίαση της έκθεσής σας. Είναι μια έκθεση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει πάρα πολλά συγκεκριμένα μέτρα και στόχους. Δεν είναι μόνο ωραία λόγια και μεγαλόστομες δηλώσεις, αλλά και πολύ συγκεκριμένοι στόχοι. Και χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τη συζήτηση. Ίσως να μην διαβάσατε ε, όλη ε, την έκθεση αυτή σε μεγάλες λεπτομέρειες. Αν θέλετε να διαβάσετε μία έκθεση του Κοινοβουλίου και να τη μελετήσετε, διαβάστε αυτή. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εγκρίθηκε και με ευρία πλειοψηφία. Ερχόμαστε λοιπόν στη συζήτηση τώρα και ελπίζω η κυρία Πιετικά να παραμείνει κατά τη διάρκεια της συζήτησης και την ευχαριστώ. Ήδη έχουν ζητήσει το λόγο πέντε συνάδελφοι. Δεν θέλω από την αρχή τη συζήτηση να επιβάλλω σκανδιναβικού χρόνου αγόρευση. Θα σας αφήσω λίγο ελεύθερου. αλλά ε, παρακαλώ έχετε υπόψη ότι δεν έχουμε ε, εδώ απεριόριστο χρόνο. Η κυρία Τόμ πρώτη, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς η Ναι, μάλιστα, τώρα ακούγομαι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι που ακούστηκε στο προηγούμενο πάνελ ρώτησε κάτι μια συνάδελφος από την Πολωνία για το ρόλο των γυναικών στα μίντια και την παρουσία τους και είπε ότι υποεκπροσωπούνται ή δεν φαίνονται αρκετά. Εγώ είμαι πρώην δημοσιογράφος και γνωρίζω πολύ καλά ότι μπορεί να ισχύει αυτό να υπάρχει μια βαθιά κρίση σήμερα, αλλά αυτό είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να ε, κάνουμε τη φωνή μας να ακούγεται πολύ περισσότερο. Δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ασφάλιση, με την παιδεία θα έρχονται όλο και περισσότερο στην επικαιρότητα. Και αυτά είναι θέματα που αφορούν τις γυναίκες και πολλές γυναίκες γνωρίζουν αυτά τα κοινωνικά ζητήματα και λιγότερο ζητήματα κρατικής ασφαλείας, ας πούμε, ενόπλων δυνάμεων. Ε, αυτό είναι απολύτως κατανοητό και θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση στις γυναίκες να ε, εκφράζονται περισσότερο, να λένε περισσότερο τις απόψεις τους για θέματα που γνωρίζουν και ε, η κρίση είναι όντως μια ευκαιρία να ακουγόμαστε περισσότερο. Άκουσα αυτά που μας είπατε τώρα και κοίταξα και πώς έχουν οι επιτροπές στη δική μας Βουλή και προς μεγάλη μου έκπληξη ε, ανακάλυψα ότι 19 γυναίκες βουλευτήνες στη Δεστονία από τις 19. Οι 9 είναι μέλη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και η Επιτροπή Εξωτερικών δεν έχει καμία, ούτε μία γυναίκα μέλος. Εμείς είμαστε λοιπόν η μόνη χώρα μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, που έχει σύνορα με τη Ρωσία. Μήπως δεν ήταν καλύτερα να έχουμε γυναίκες να διαπραγματεύονται αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μαρατίδου, παρακαλώ, από την Ελλάδα. Ε, σας ευχαριστώ για δεύτερη φορά. Ε, ε ήταν, πολύ, ήταν εξαιρετική η παρουσία ε, που μας έγινε για αυτήν την έκθεση. Ε, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων προσπάθησε να καλύψει τις διαφορές μεταξύ ανδρών γυναικών στην αποσχόληση, στην εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία με την, βέβαια, με την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ε, συμβεί κιόλα. Στα εθνικά κοινοβούλια έχουμε σοβαρά τα προβλήματα. Βέβαια, από την πρωινή συναντρίαση είδαμε όντως ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ε, το τελευταίο διάστημα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες πρώτα απ' όλα στην αγορά εργασίας περισσότερες γυναίκες στις διαδικασίες ύψης ε, πολιτικών αποφάσεων και αναγνωρίζουμε όμως ότι ο συνδυασμός της οικογενειακής ε, και επαγγελματική ζωή είναι καθοριστική σημασία για την ίση συμμετοχή ε, στην αγορά εργασία. Από εκεί ξεκινάει για να μπορέσουμε να πάμε στο, σε δεύτερο επίπεδο στην πολιτική και το λέω ε, εγώ η οποία ε, προέρχομαι από, ε, μια χώρα η οποία είναι πατριαρχική γιατί υπόθηκε πιο μπροστά στη συζήτηση είμαι παντρεμένη, έχω τρία παιδιά ε, να το πω έτσι χαριτολογώντας την ε, συνάδελφο από την Εστονία που ο άντρας μου δεν, είπε, δεν μου είπε να διαλέξω ένα από τα δύο γιατί ίσως πιο μπροστά είχα κατακτήσει προσωπικά έναν άλλον χώρο που ήταν κατεξοχήν ανδρικός τα γεωργικά μηχανήματα διότι ασχολούμαι ε, στη δουλειά, η δουλειά μου ήταν αυτή εμπόριο με γεωργικά μηχανήματα καταλαβαίνετε ότι μέσα από την, αγορά, μέσα από την εργασία κατακτήθηκε και το άλλο το κομμάτι τουλάχιστον στην δική μου την περίπτωση. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν... Ε, ε, να σας δώσω μάλλον και κάποια ακόμη στοιχεία είχα δώσει κάποια πιο μπροστά για τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται και είναι υψηλότερα τα ποσοστά των γυναικών μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο χωρίς βεβαίως να πούμε ότι τα ποσοστά στην κυβέρνηση στο προεδρείο της βουλής ή οι γυναίκες που συμμετέχουν ως ε, βουλευτίνες ε, στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι ε, αντίστοιχο. Έχουμε μόνο δύο γυναίκες στην κυβέρνηση, έχουμε μία γυναίκα αντιπρόεδρο πρόεδρο στην ε, Ελληνική Βουλή και 63 όπως είχα πει το πρωί στους 300 που είμαστε γυναίκες. Ε, η κυρία Άννη Ποδηματά είναι μία από τις 7 γυναίκες ε, της ευρωομάδας, της ελληνικής ευρωομάδας που αποτελείται από 22 ευρωβουλευτές και εκεί έχουμε μια εκπροσώπηση που θα μπορούσε να ήταν πολύ, είναι ακριβώς στην ποσόστοση μπορώ να πω ε, και θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη και όσον αφορά τώρα τα κόμματα ε, θα πρέπει να υπάρξει η συμμετοχή πρώτα απ' όλα ως κομματικά μέλη στα κόμματα γιατί έτσι είναι δομημένη η δημοκρατία ε, μέσα στα κόμματα και να μπορούν μέσα από τα κόμματα να είναι σε θέσεις ευθύνης. Από εκεί ξεκινάει. Ε, θέλω να πω ότι η οικονομική κρίση που είναι μια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος πλήττει ακόμη περισσότερο τις γυναίκες και ακριβώς ε, ε, επειδή αυτό είναι ε, μία αναφορά που ε, την έχετε κάνει και εσείς και θα το δείτε και ως ε, μία συνάντηση γυναίκα και οικονομική κρίση, μάλλον οικονομική κρίση και γυναίκα. Θέλω να πω ότι με έκπληξη να σας μεταφέρω κάτι που συνέβη την τελευταία εβδομάδα στην ε, Ελλάδα με έκπληξη διαβάσαμε στον τύπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα καταργηθεί το μέτρο της ποσόστοση για τη συμμετοχή των δύο φύλων στα υπηρεσιακά ε, συμβούλια των δημόσιων υπηρεσιών, δηλαδή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ε, δημοσίου δικαίου όπως θα αναφέρουμε εμείς στη χώρα μας. Ε, τα οποία είχαν εισηγηθεί με έναν νόμο το 2000 δηλαδή θα κάνουμε πίσω σε κατακτήσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Ε, το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. Εμείς θα θέλουμε πολύ μεγαλύτερη ε, συμμετοχή και επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι ε, ελάχιστος και θα πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι ε, συνάδελφοι και συναδέλφισες ε, θέλω να ευχαριστήσω και να μεταφέρω από την Ελλάδα ένα μήνυμα αισιοδοξία προς τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς, ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου, ότι οι Έλληνες ε, είμαστε αυτοί που στεκόμαστε στα πόδια μας παρόλο ότι έχουμε κατασυγκοφαντηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα το έλεγα στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά ο χρόνος δεν μου το επέτρεπε και ε, στο τέλος θα ήθελα να πω κάτι που βλέπω μέσα εδώ στο, σε αυτή την αίθουσα που είμαστε ε, αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και μεταφέρουν τη δική μας φωνή στα αυτιά όλων σε όλες τις γλώσσες που αποτελούμε ε, αυτήν την ε, συνάντηση σήμερα, στους διερμηνείς που είναι στις καμπίνες και αυτό που βλέπω είναι ότι θα πρέπει μάλλον να μπει μια ποσόστοση υπέρ των ανδρών διότι εδώ είναι πραγματικά η κατάκτηση είναι των γυναικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα αρχίζουν οι σκανδιναβικοί χρόνοι αγόρευσης, όπως σας είχα ανακοινώσει προηγουμένως. λοιπόν, βάζω όριο. Τρίλεπτο. Έκαστος. Γιατί έχουμε πολλούς εγγεγραμμένους και δεν θα προκάνουμε. Πρέπει να απαντήσει και η κυρία Πιετικάινεν. Ε, παρακαλώ, ε, τρίλεπτο καθένας. Η κυρία Χτέν από την Τουρκία, παρακαλώ. Yes. Uh, I am also the member of the... Uh, Και εγώ θα ήθελα. Επίσης, εγώ θέλω να μιλήσω για την παιδεία τον πολιτισμό και την νεότητα και είμαι υπεύθυνη κιόλας για αυτά στο Κοινοβούλιο, για αυτά τα θέματα. Στη χώρα μου, την Τουρκία, το, η τελευταία συνταγματική τροποποίηση που βασίζεται στο δημοψήφισμα του 12 Σεπτεμβρίου 2010 ε, ενίσχυσε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών εισάγοντας τη θετική, τις θετικές διακρίσεις για ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ανάπηροι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε λοιπόν στενές σχέσεις με όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Όμως, γιατί αυτές οι ομάδες όσο λιγότερο είναι ε, εκπαιδευμένες, τόσο πιο ευάλωτες είναι. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην παιδεία για να μπορούν να φτάσουν στη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Έχουμε πολλές ανισότητες ε, στην ε, Τουρκία και ξεκινάμε ε, εθνική εκστρατεία όπου συμμετέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμα και ο ιδιωτικός τομέας. Αυτές είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις και έχουν επηρεάσει και τη βασική εκπαίδευση όπου το ποσοστό παρακολούθησης του δημοτικού είναι 96% ενώ είναι μόλις 82% για τα κορίτσια. Θέλουμε να λύσουμε και το πρόβλημα του αλφαβητισμού των ενήλικων γυναικών. Έχουμε Πολλά εκατομμύρια τελείως απέδευτες και αναλφάβητες γυναίκες στην ηλικία των 50 και άνω. φτιάχνονται ειδικά βιβλία και, εκπαιδευτικά, ε, και εκπαιδευτικό υλικό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στον αλφαβητισμό των γυναικών. Στο Κοινοβούλιο εμείς έχουμε σχετική νομοθεσία και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα επιτεύγματά μας όσον αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την, της ισότητας των φύλων. Στις 8 Μαρτίου 2012 εμείς εγκρίναμε την νομοθεσία για την προστασία της οικογένειας και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Είχαμε τέσσερα άρθρα σε αυτή την νομοθεσία και τελικά της δώσαμε περισσότερη ουσία επεκτείνοντας τη σχετική, την νομοθεσία αυτή σε 25 άρθρα. Οι γυναίκες ε, είναι σημαντικές και φροντίζουν για όλα τα άλλα τα μέλη της οικογένειας και γι' αυτό θέλουμε και έχουμε καλύψει όλες τις πτυχές ε, της δικαστικής διαδικασίας. Ε, μπορείτε να μου δώσετε άλλο ένα λεπτό παρακαλώ. Oh, okay, it's problem because I... Όχι, έχω πρόβλημα, γιατί άμα ο καθένας πάρει ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι, ναι, γι' αυτό σας ζήτησα άλλο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας. Ε, εμείς έχουμε για πρώτη φορά ε, επιδόματα ε, παιδιών για τις ε, γυναίκες που εργάζονται και στην περίπτωση που η γυναίκα χάσει το 10% της δυνατότητας προσεργασία θεωρείται ήδη ανάπηρη. Και Επίσης, καταβάλλεται το 10, η σύνταξη της ε, τυχόν αποθανούσας μητέρας ε, στα παιδιά ή στους ε, όσους ε, εκείνη είχε αναλάβει. Επίσης στις βιομηχανικές ζώνες όπου οι γυναίκες εργάζονται πάρα πολύ εντατικά και σκληρά, η ασφάλισή τους είναι πολύ πιο σημαντική, το ίδιο και για τους γεωργούς. Κοινωνική πρόνοια υπάρχει επίσης για τις άνεργες γυναίκες και έχουμε αυξήσει τη συμμετοχή ε, των γυναικών μας ε, στο εργατικό δυναμικό από το 23% στο 28%. Στην Τουρκία δίνουμε μεγάλη σημασία στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και στο διεθνές επίπεδο. Μια από τις πιο δυναμικές οικονομίες του κόσμου, ως ευρωπαϊκή χώρα, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και υποψήφια χώρα στην Ένωση, θα ήθελα να επαναλάβω τη βούλησή μας να συνεργαστούμε με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και με τα κοινοβούλια των κρατών μελών για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά μου φάγατε. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Βόντα από την Σλοβενία. Ευχαριστώ πολύ. Στο Σλοβενικό Κοινοβούλιο οι πρόσφατες εκλογές ήταν το 2011 και το 1 τρίτο των βουλευτών ήταν γυναίκες και 40% των πρόεδρων των διαφορετικών φορέων στο Σλοβενικό Κοινοβούλιο είναι γυναίκες. Έχουμε κάνει κάποια πρόοδο, έχουμε ακόμα όμως πολλά να πετύχουμε γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχει μόνο μία γυναίκα. Και δεν έχει χαρτοφυλάκιο κιόλα αυτή η Υπουργό. Είναι αυτά τα οποία ανέφερε προηγουμένω η κυρία Πιέτη κάνει γιατί τον διαχωρισμό των θέσεων εξουσία. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, ξέρουμε πόσο απέχουμε από την πραγματική ισότητα. Πολλές φορές βλέπουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις ότι το υποσυνείδητο γίνεται συνειδητό, αν μου επιτρέψετε να το πω έτσι, ότι αταβιστικές και υποσυνείδητες μορφές αντίληψης έρχονται στην επιφάνεια και αυτό είναι ένα στοιχείο που προσδιορίζει και τους κοινωνικούς ρόλους μας. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν υποδέστερη θέση στην πολιτική, όπως και γενικά. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για κάτι τέτοιο συγκεκριμένα. Οι γυναίκες πολλές φορές θέτουν ερωτήματα τα οποία οφείλονται στο γεγονός ότι οι γυναίκες συνήθως έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλούς ρόλους στην ε, κοινωνία και συγχρόνως οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να αντιπα να αντιπαρατίθενται σε στερεότυπα και σε προκατηλημένες απόψεις από την πλευρά των ανδρών. Μας κολλάνε ετικέτες, ρετσέτες, στερεότυπα που έχουν να κάνουν με το γυναικείο φύλλο. Συμπεριφορές που υποτίθεται ότι είναι γυναικείες, θηλυκές. Οι άντρες ξέρουν ότι όλα αυτά δεν αληθεύουν, αλλά μέσα στο πολιτικό παιχνίδι χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτό το όπλο. Υπάρχει και κάτι τρίτο το οποίο και αυτό είναι πολύ προβληματικό. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές κοινωνίες σε αυτή την αίθουσα και ξέρω ότι είναι διαφορετικές οι κοινωνίες μας, αλλά στη δική μας χώρα, στη Σλοβενία, υπάρχουν πολλές φορές έντονες κριτικές από γυναίκες προς την κατεύθυνση άλλων γυναικών. Πολλές φορές οι γυναίκες είναι αυτές που επικρίνουν τις άλλες γυναίκες και δεν συνειδητοποιούν ότι από τη μία πλευρά είναι θύματα αλλά και θύτες. Και είναι αυτές ακριβώς οι οποίες πολλές φορές διατηρούν και διαιωνίζουν τις προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών. Νομίζω ότι στην εκθεσή σας αναφέρατε μια πλευρα ειναι θυματα αλλα και θυτες και ειναι αυτες ακριβως οι οποιες πολλες φορες διατηρουν και διαιωνιζουν τις προκαταληψεις σε των γυναικων νομιζω οτι στην εκθεση σας αναφερατε μια λυση και η λύση είναι να βοηθήσουμε τις γυναίκες να διαδικτυωθούν περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ τους, όχι μονάχα σε ένα κράτος, σε μια κοινωνία, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Θα προσπαθήσω να, μείνω εντό του χρονικού όριου που μου δώσατε. Ήθελα να πω ότι αυτή η συνεδρίαση γίνεται σε μια φάση πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, όπου συζητάτε το μέλλον τη Ευρώπη. Και όλοι εμά και κυρίω οι χώρε που αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερε δυσκολίε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να φτιαχτούν ε, οι Ηνωμένε τη Ευρώπη χωρί τον Νότο της Ευρώπης και χωρίς ε, το όσους υπόκειται σε διακρίσεις, χωρίς τις γυναίκες και χωρίς τους νέους. Για να μιλήσω για την Ιταλία, ήθελα να πω ότι η κατάσταση στην Ιταλία πιθανότητα είναι γνωστή. Εμείς ε, από το 2008 ε, έχουμε προχωρήσει πολύ. Ήμασταν 138 γυναίκες, στη Γερουσία 58. Είμαστε περίπου στο 21,43% γυναικών. Μόνο μία η Λέδη Μονταλτσίνη είναι γερουσιαστής ε, διαβίου και είναι και εκείνη που έχει κερδίσει το βραβείο Νόμπελ. Δεν είμαστε σε πολύ ικανοποιητικά ποσοστά λοιπόν. Ήθελα επίσης να πω ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχει Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών από το 2000 ε, και έχει αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες γιατί τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ αλλά σίγουρα έχουν αλλάξει λόγω των συνθηκών ζωής. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Επτά γυναίκες βουλευτές απέκτησαν παιδί αυτή τη θητεία. Νέες βουλευτίνες και άλλαξε η κατάσταση είχαν ε, άδεια ε, εγκυμοσύνης γονική άδεια. Υπάρχει λοιπόν εξέλιξη όχι μόνο στους θεσμούς αλλά και στη χώρα μας. Θα έχετε ακούσει και για εκείνο το φαινόμενο αν δεν γίνει τώρα πότε ε, και δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο, αλλά είναι και πολιτικό φαινόμενο και έχει εξαπλωθεί σε διάφορες χώρες της Ένωσης και μας έχει εγκαλέσει στις δραστηριότητές μας στο Κοινοβούλιο. Η συνάδελφος ανέφερε την κοινωνία που προβλέπει την ε, ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για άλλες προτάσεις που σίγουρα βοηθήθηκαν από τον εξωτερικό κόσμο, από τον κόσμο των γυναικών που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία. Ε, έχω Έχει να κάνει με μια νομοθεσία που εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τη Γερουσία και πρόκειται ε, για τις γυναίκες που εκλέγονται στους Δήμους και στις τοπικές αρχές και έχει να κάνει και με τους διαγωνισμούς. Ε, σκεφτήκαμε πως ήταν πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από τις τοπικές αρχές για να σεβαστούμε την ισότητα των φύλων. Ίσως θα πρέπει να το καταλάβουμε και στην Ευρώπη ότι αν δεν ξεκινήσουμε από το χαμηλότερο επίπεδο δεν θα τα καταφέρουμε. Μια άλλη νομοθεσία αφορά τη χρηματοδότηση των κομμάτων και ένα κομμάτι της χρηματοδότησης αφαιρείται αν ως κύρωση δηλαδή, ως ποινή για τα κόμματα που δεν σέβονται ε, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών που πρέπει. Πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν μια ποιότητα στην πολιτική και στο διοικητικό μηχανισμό. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρώπη είναι να επηρεάσει τα χρονοδιαγράμματα, γιατί μεγάλο κομμάτι τη νομοθεσία που περνά από το Ιταλικό Κοινοβούλιο εξαρτάται και προωθείται από την Ευρώπη. Θα πρέπει να βοηθηθούν λοιπόν τα πολιτικά κόμματα να λάβουν ε, τι ευθύνε του. Να σα πω ότι συζητείται αυτή τη στιγμή ένα, μια νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα, άρθρο 48 του συντάγματο. Θα πρέπει να κάνει και η Ευρώπη τη δική τη προσπάθεια όπως έκανε για τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό, τη διαφθόρα και για το πρόβλημα των γυναικών, γιατί πιστεύω ότι έχουν πολλά να γίνουν ακόμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Πόντος Ταμιάσκα από την Πολωνία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Είμαι γερουσιαστής και εργάζομαι στην Επιτροπή Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι σημαντικά τα χειρήματα που έχει αναλάβει η Βουλή και η Γερουσία στην Πολωνία για να προωθηθεί η γυναικεία παρουσία στα κοινά. Το 2011 εγκρίθηκε νόμος που τροποποιεί τον εκλογικό νόμο στη χώρα και αφορά την ε, ισομερή εκπροσώπηση στα ψηφοδέλτια. Από το 2011 τίθεται σε ισχύ, είναι σημαντικές οι πρόνοιες και οι διατάξεις. Στο ε, ψηφοδέλτιο λοιπόν για τη Βουλή μας, ΣΕΙΜ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η συμμετοχή ανδρών και γυναικών ρυθμίζεται δια νόμου και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% για κάθε φύλλο. Στη συνέχεια, η κύρωση που υφίστανται τα κόμματα είναι να μην ε, γίνει δεκτή επίσημα μια λίστα τους και ε, σε ό,τι αφορά τις εκλογές του 2011 και το αποτέλεσμά του, η Βουλή μας απαρτίζεται κατά 24% από γυναίκες. Στην προηγούμενη θητεία το ποσοστό αυτό ήταν 20% και στη Γερουσία είναι 12% σήμερα. Η πρόεδρος της Βουλής είναι γυναίκα για πρώτη φορά στην ιστορία της Πολωνίας. Άλλο σημαντικός νόμος που εγκρίναμε αφορούσε την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και εντός οικογένειας. Η ε, Πολωνική Βουλή ε, ενημέρωσε το 2009 το σχετικό νόμο και με τις αλλαγές που έγιναν και ε, δημιουργήθηκε μάλλον ένα πρόγραμμα για την πρόληψη της βίας στην οικογένεια. Αυτό δράσε όλα τα επίπεδα ε, της ε, διοίκησης με συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία για να ε, αποφεύγεται και να αποτρέπεται η βία στην οικογένεια. Το 2009 αποφάσισε η Βουλή μας να προσυπογράψει μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της βίας στην οικογένεια ε, της ενδοοικογενειακής βίας. Γνωρίζουμε ότι ε, άλλα 12 κράτη-μέλη την έχουν υπογράψει. Εμείς ε, πρόκειται να την υπογράψουμε για να γίνει δεκτή αυτή η αλλαγή η οποία υπευλήθη από την πλατφόρμα των πολιτών που είναι το κυβερνών κόμμα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά το ζήτημα του βιασμού και της ε, ποινική δίωξης του βιασμού. Μέχρι σήμερα τι ισχύει στην Πολωνία. Έπρεπε το θύμα να συμφωνήσει για να αρχίσει η ποινική δίωξη του δράστη. Δυστυχώς αυτό ανάγεται ως νομοθεσία στο 1932 και είχε στόχο να αποτρέψει τη διαπόμπευση δημοσίως των θυμάτων βιασμού. Τώρα Δηλαδή μέχρι τώρα δεν μπορούσε να κινήσει η ποινική δίωξη ε, αν δεν έδινε τη συγκατάθεσή του το θύμα. Τώρα γίνεται αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα. Ε, και... Ε, ο άλλος νόμος που ψηφίστηκε αφορά την ημερήσια φροντίδα των παιδιών ηλικίας άνω των τριών ετών. Βρεφών σταθμή και αντίστοιχες δομές, νηπιαγωγία, ε, αυτά τα ιδρύματα δεν θα θεωρούνται νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά εκπαιδευτικά πλέον. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα, διάφορα είδη ε, φύλαξης παιδιών και εκτός από τους βρεφονηπιακούς και ε, τα νηπιαγωγεία υπάρχουν και ατομικές ε, υπηρεσίες που παρέχονται από babysitter, από γυναίκες που κρατούν παιδιά και ε, πληρώνονται από το σύστημα υγείας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα ε, και ε, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Θέλω να προσθέσω ότι κάθε χρόνο διοργανώνουμε στην Πολωνία ένα συνέδριο γυναικών και κερδίζει και σε δημοφιλία και μεταξύ των ε, πολιτικών. Ήρθε και ο πρόεδρος φέτος και ο Πρωθυπουργό και μάλιστα έχει και διεθνή παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο χρόνος τελειώνει. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Σουηδίας. Στην Σουηδία έχουμε σχεδόν ισότητα των φίλων στο Κοινοβούλιο και στην ε, κυβέρνηση. Και ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι ότι έχουμε πολύ καλή πρόνοια για τα παιδιά και γονική άδεια προβλέπεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι γυναίκες να μπορούν να δουλεύουν ε, και να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Υπάρχουν διάφορα πολιτικά κόμματα που φτιάχνουν τις λίστες τους με τέτοιο τρόπο, τους εκλογικού καταλόγους, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 50-50 γυναίκες άντρες. Και αυτό ενθάρρυνε και άλλα πολιτικά κόμματα να βάλουν περισσότερες γυναίκες στα, τους, στα ψηφοδέλτιά τους. Είναι δυνατόν να συνδυάσει κανείς την πολιτική εργασία και δραστηριότητα με την γονική ζωή, με την ε, οικογενειακή ζωή, γιατί έχουμε ένα σωρό εβδομάδε που δεν υπάρχει ολομέλεια και υπάρχει και ομάδα αναφοράς όπου υπάρχουν γυναίκες από διάφορες πολιτικές ομάδες, από τα διάφορα πολιτικά κόμματα και εκεί συζητάμε τι τυχόν δεν πάει καλά, οργανώνουμε σεμινάρια, ειδική κατάρτιση, ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε, να δουλέψουμε καλύτερα μέσα σε ένα πλαίσιο ισότητας των φύλων. Για τα μέλη του Ισοειδικού Κοινοβουλίου, όταν, ε, όπου έχουμε τη δυνατότητα για πρόνοια για τα παιδιά όταν, όσο εργαζόμαστε μέσα στο κοινοβούλιο μπορούμε επίσης να πάρουμε γονική άδεια σημαίνει ότι έρχεται κάποιος αντικαταστάτης, κάποιος αναπληρωτής για την περίοδο όπου έχεις τη γονική άδεια. Μάλιστα είναι το επόμενο άτομο που βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματός σας, του κόμματός σου που έρχεται και σε αντικαθιστά όσο δεν μπορείς εσύ. Κάτι ακόμα που έχουμε στη Σουηδία είναι ότι δεν έχουμε μόνο μία Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, αλλά αυτή αποτελεί κομμάτι της Επιτροπής Απασχόλησης και όλα τα θέματα ισότητας των φύλων δεν τα εξετάζει απλά αυτή η Επιτροπή, αλλά περνούν και μέσα από όλες τις Επιτροπές. η ιδέα είναι δηλαδή ότι κάθε κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τις πολιτικές μέσα από την οπτική της ισότητας των φύλων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι γυναίκες και άνδρες είναι γονείς και οι γυναίκες και άνδρες χρειάζεται να μοιράζονται τις ευθύνες. Και ε, να έχουν τα δικαιώματα να εργάζονται και να κερδίζουν ε, τη ζωή τους αλλά και να συμμετέχουν πολιτικά αλλά να έχουν και το δικαίωμα σε σταδιοδρομία. Τελευταίος ομιλητής πριν από την κυρία Πιετικάινεν που θα κλείσει αυτό το πάνελ Τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Λάβισκ από τη Γερμανία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομη αλλά ήθελα να περιορίσω αυτά τα οποία θα πω σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, στο βασικό νόμο της Γερμανίας, που έχει συνταγματικό χαρακτήρα, έχουμε τονίσει ότι ένας από τους στόχους του συντάγματος είναι η ισότητα των ανδρών και των γυναικών. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εμείς ως βουλευτές δεν το δεν αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε όσο θα έπρεπε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία άκουσα από τους διάφορους συνάδελφους και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τονίσουμε στην Γερμανική Βουλή ότι θα πρέπει να εξυπηρετείται ο στόχος αυτός της ισότητας ανδρών και γυναικών και να είμαστε λίγο πιο ενεργοί για τα θέματα αυτά. Έχουμε πάρει πρόσφατα μια έκθεση για την σύνθεση των διαφόρων αξιωμάτων και φορέων στην ε, Γερμανία. Και εκεί μπορεί να υπάρξει και κάποια επιρροή των βουλευτών της Bundestag σε σχέση με τη σύνθεση αυτών των φορέων. Παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο ασχολείται με την υγεία των γυναικών και των παιδιών και όπου δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Εδώ είναι φανερό ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις. Πολλές φορές είναι αυτά λεπτομεριακά θέματα, αλλά αυτά σας κάνουν πιο σαφή και την εικόνα. Και νομίζω ότι δείχνουν ότι θα πρέπει να δράσουμε και σε χώρους οι οποίοι δεν είναι τόσο ορατοί όσο ο πολιτικός χώρος αν θέλουμε πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πραγματικά μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και θα εξασφαλιστεί ότι θα λαμβάνει ο κόσμος στα σοβαρά και την ε, πολιτική ισότητα που είναι πράγματι μια συνταγματική επιταγή για τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δίνω λόγο στην κυρία Πιετικάινεν για να απαντήσει στα διάφορα σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για όλα τα σχόλια που έχετε διατυπώσει. Μερικές παρατηρήσεις ε, μονάχα. Ναι, κατανοώ αυτό που είπατε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει η λεγόμενη επιστροφή του μαστιγίου ότι τα πράγματα οδηγούν στο να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση κατά των γυναικών και να οξύνεται ακόμα περισσότερο η ανισότητα. Και πράγματι αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα ότι η περιθωρικοποίηση πλήττει πολύ πιο συχνά τις γυναίκες, ιδίως τα κράτη-μέλη, τα οποία τώρα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και αυτό θα πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Επίσης, τρίτον, και το θέμα των μέσων ενημέρωσης και εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Και τέταρτον, η δυνατότητα των κυρώσεων. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε μέσα στα πλαίσια της εξέτασης των βελτίστων πρακτικών στις ε, χώρες μέρες μας. Και ακούμε, ακούσαμε πολλά για αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε περισσότερο, να ανταλλάξουμε απόψεις και βέλτιστες πρακτικές. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και αν σας ενδιαφέρει μπορείτε από τη στιγμή που θα γυρίσετε στις πατρίδες σας και θα συζητήσετε με τους συναδέλφους σας και τις συναδέλφους σας εάν ενδιαφέρεστε να έχετε μια πιο ε, τακτική άτυπη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Ελπίζω να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για να εκδηλώσετε την πρόθεσή σας. Νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος μου, τελείωσε πράγματι, είναι 3,5. Αλλά μου υποσχέθηκε ο πρόεδρος και δύο-τρία λεπτά ακόμα. Αυτό το οποίο νομίζω θα ήταν σημαντικό εν ώψη του μέλλοντος είναι το θέμα της καλύτερης συνεργασίας μας στο μέλλον. Ξέρετε ότι έχουμε τη συνεδρία της ΚΟΣΑΚ, συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια που είναι πολύ χρήσιμες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επαρκείς αυτές οι συνεδριάσεις και δεν είναι πάντα δυνατό για όλες μας να ταξιδεύουμε εμείς στις χώρες σας ή εσείς στις Βρυξέλλες. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να βρούμε και ένα άλλο παράλληλο τρόπο για να συνεργαζόμαστε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίζουμε περισσότερο τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συνάδελφοί μας σε διάφορα κράτη-μέλη. Η πρόταση αυτή της εκστρατείας 50-50, 50%-50% είναι μια εκστρατεία που νομίζω ότι μπορεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν σας ενδιαφέρει και εσάς και ποιες είναι οι αντιδράσεις σας. Αν έχω λοιπόν λίγο ακόμα χρόνο, ίσως θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στο θέμα των μέσων ενημέρωσης, γιατί και αυτό συνδέεται με την αρνητική αντίδραση που έχει υπάρξει κατά των γυναικών λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς με νομοθετικά μέτρα ή οποιαδήποτε δράση. Είναι μόνο σε προσωπικό επίπεδο και το πώς εμείς παρουσιάζουμε και υπερασπιζόμαστε τις γυναίκες και το ρόλο των γυναικών στην πολιτική και πώς παρουσιάζουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανισότητα που θα παίξει ρόλο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα μονάχα για αυτό το θέμα. Για όλη αυτή τη συζήτηση για τις ποσοστώσεις. Και σίγουρα θα ακούσουμε και περισσότερα για το θέμα αυτό όταν έρθει η Επίτροπος Ρέντινγκ εγώ πραγματικά στενοχωριέμαι πολύ όταν μου λένε γυναίκες ε, συνάδελφοι, ανεξάρτητα από αυτό που πιστεύουν για τις ποσοστώσεις, ότι προτιμώ να μην παρέμβω ε, στο θέμα αυτό και μου λένε ότι δεν είναι καλή ιδέα οι ποσοστώσεις γιατί θα πρέπει να διαλέγουμε μόνο τους καλύτερους, τις καλύτερες και να μην υπάρχει υποστήριξη. Επομένως, στι ποσοστώσει. Μα εγώ δεν κατάλαβα κανεί να υποστηρίζει ποσοστώσει λέγοντα να εκλέγουμε άσχετε γυναίκε. Και όντα γυναίκα, νο, να λέει κάποιο ότι εγώ θέλω να εκλέγομαι μόνο λόγω της ε, αξίας μου, είναι σαν να λέει ότι κανονικά μια γυναίκα δεν έχει την αξία αυτή σε αξιοκρατικό σύστημα, δεν θα εκλεγόταν. Εγώ λέω στους συναδέλφους μου, βρίσκομαι εδώ γιατί έχω κάποια αξία. Και εσείς πάλι που υποστηρίζετε τις ποσοστώσεις και εσείς το κάνετε γιατί. Γιατί δεν είσαστε ικανοί. Δηλαδή είναι ένα, μια αντιμετώπιση ότι μόνο ότι οι μόνες γυναίκες που υποστηρίζουν τις ποσοστώσεις είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν αξία. Και δεν νομίζω ότι οι γυναίκε αυτέ που στρέφονται κατά των ποσοστώσεων σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά αθέλητά μα πάρα πολλέ φορέ εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα. Ότι κάπου παίρνουμε σαν δεδομένο ότι οι γυναίκες είναι χαμηλότερες ποιότητας και ότι είναι σαν να δίνουμε την εντύπωση ότι δεν είναι λογικό ή είναι δίκαιο ή είναι αδικαιολόγητο το να επιβάλλουμε τις ποσοστώσεις. Αυτή την εντύπωση δημιουργούμε οι ίδιες πολλές φορές. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς θέτουμε αυτά τα ζητήματα, πώς τα συζητούμε, πώς τα παρουσιάζουμε μαζί με τις γυναίκες συναδέλφους μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δύο ακόμα μικρά πράγματα όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε τα ζητήματά μας. Αν μπορείτε να παραθέσετε αυτά που είπε μια γυναίκα, αν μπορείτε να κάνετε μια αναφορά σε μια γυναίκα, αν μπορείτε να επενέσετε μια άλλη γυναίκα, δεν χάνετε εσείς τίποτα. Αλλά αυτό δείχνει ότι μια άλλη γυναίκα μπορεί πράγματι να προτείνει κάτι καλό, να πει μια έξυπνη να κάνει κάτι σημαντικό. Και όταν εγώ μπορώ πάντα να εξάρω το έργο μιας γυναίκας και αν μπορώ να συνδέσω μια έξυπνη γυναίκα με μια άλλη έξυπνη γυναίκα ή έστω και με ένα έξυπνο άνδρα, αυτό δεν καταδαπανά το χρόνο μου και δεν χάνω εγώ προσωπικά τίποτα. Αλλά με τον τρόπο αυτό βοηθάτε, βάζετε ένα μικρό πετραδάκι που θα βοηθήσει ίσως μια άλλη γυναίκα στις προσπάθειές της να πετύχει τους πολιτικούς στόχους και την ισότητα που διεκδικούμε και πιστεύω πραγματικά ότι όταν επενούμε ως γυναίκες τις άλλες γυναίκες, όταν συνεργαζόμαστε και όταν τις βοηθούμε να επιτύχουν αυτά που θέλουν σε καθημερινό επίπεδο, μπορούμε να διευκολύνουμε το έργο όλων μας. Και μπορούμε επίσης να δώσουμε και ένα καλό παράδειγμα για τις νεαρές κοπέλες ότι το να είναι για να είναι κανείς γυναίκα είναι σημαντικό και το να είναι πρωθυπουργό ή πρόεδρος μια γυναίκα είναι όχι μόνο φυσιολογικό αλλά και πολύ θετικό και ότι μπορούν και τα νέα κορίτσια να ονειρεύονται να καταλάβουν αυτές τις θέσεις όταν μεγαλώσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πιετικάινεν για αυτά τα συμπεράσματα. Με μεγάλη χαρά είδαμε αυτή τη συζήτηση και ακούσαμε πάρα πολλά σημαντικά σχόλια που μας περιγράφουν την κατάσταση και στα διάφορα κράτη-μέλη. Και ε, θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω δύο πράγματα. Ακούμε όλο και περισσότερο θα πρέπει να έχουν περισσότερη εξουσία στην πολιτική οι γυναίκες και αυτό τι σημαίνει, θα πρέπει να παραιτηθούν οι άντρε να κάνουν ένα βήμα πίσω. Ναι, ακριβώ. Αυτό θα πρέπει να κάνουν οι άντρε, ένα βήμα πίσω για να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία γυναίκε. Γιατί μέχρι τώρα τη μερίδα του λέοντο την έχουν οι άντρε. Βεβαίω να υποχωρήσουν λίγο για να προωθηθούν οι γυναίκες. Και για τις ποσοστώσεις, το είπαν και οι κυρίες Πιετικάινεν και Αντζελίλη, και εγώ χτες είχα την ευκαιρία να πω ότι οι ποσοστώσεις μπορεί να μην είναι το υπαριθμόν ένα μέσο και εργαλείο, αλλά είναι ένα μέσο αποτελεσματικό για να επιτύχουμε κάτι, γιατί πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν κάποιος αρνείται την ποσόστοση, αυτό τι σημαίνει. Ότι η εναλλακτική λύση είναι να αλλάξει το ισχύον σύστημα, γιατί μέχρι τώρα έχουμε ποσοστώσεις υπέρ των ανδρών. Δηλαδή, με άτυπε βέβαια ποσοστώσει προωθούνται οι άνδρες. Οι άνδρες προ... Ε, εκλέγουν άνδρες. Οι άνδρες διορίζουν άνδρες. Ε, αυτή είναι η ποσόστοση και η πρόθεση των ανδρών. Και μάλιστα είναι άτυπη και αφανής. Δεν υπάρχει επίσημη ποσόστοση, αλλά στην πράξη αυτό ισχύει. Ακριβώς όπως είπε και η κυρία Πιετικάινεν, και εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει ότι οι γυναίκε δεν έχουν τα προσόντα και βέβαια τα έχουν. Αλλά οι άνδρες ελέγχουν την εξουσία και έτσι επιβάλλουν την ποσόστοσή του με τρόπο σκοτεινό και αόρατο. Θα πρέπει λοιπόν να σπάσει αυτό το σύστημα για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι γυναίκες. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους ε, θερμά για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Προσπαθώ λίγο να κερδίσω χρόνο μέχρι να έρθει η κυρία Ρέντινγκ επάνω εδώ στο πάνελ. Eh, Μάλιστα. Λοιπόν, είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή η ευκαιρία που έχω εδώ να καλωσορίζω την κυρία Ρέντινγκ, την Επίτροπο. Ε, καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο και βρήκατε το χρόνο να έρθετε να συζητήσετε μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας και περιμένουμε να ακούσουμε την τοποθέτησή σας. Πριν σας δώσω το λόγο, κυρία Ρέντινγκ, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντζελίλη που έχει να κάνει μια ανακοίνωση, μια δήλωση και μετά η Επίτροπος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί είχαμε δύο μέρες πολύ εντατικές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ μάλλον από καρδιά στην Επίτροπο Ρέντινγκ που βρήκε το χρόνο να έρθει σήμερα εδώ μαζί μας. Βίβιαν, εγώ δεν θα σου ανακεφαλαιώσω τα νούμερα και τα στοιχεία, γιατί εσύ τα γνωρίζεις όπως και εμείς και καλύτερα από εμά. Θα ήθελα μόνο να σου πω δύο πράγματα. Δηλαδή, από αυτό, αυτή τη διάσκεψη και από τη σημερινή συζήτηση προέκυψε ένας στόχος ότι δηλαδή οι θεσμοί θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν και μετά στο εσωτερικό, στις ευρωπαϊκές δηλαδή καταστάσεις να υπάρχει αντικειμενικά ανισότητα όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα. Μπορούμε να δώσουμε το παράδειγμα το λαμπρό της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο, να πούμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο δύο, από τις 20, από, μόνο δύο γυναίκες ήταν πρόεδροι του Κοινοβουλίου από 29. Μπορούμε να πούμε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος της Κομισιόν γυναίκα. Μπορώ να συνεχίσω και να πω και άλλα παραδείγματα, αλλά τα, στοιχεία αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι πρέπει εμείς να δίνουμε το, το σωστό παράδειγμα και έπειτα είμαστε έτοιμες να σε στηρίξουμε για τον αγώνα για τις ποσοστώσει. διότι θεωρούμε, και το έλεγε και ο πρόεδρο μόλι, ο πρόεδρο Γκούσταυσον, ότι στόχος μας είναι να αλλάξει το σύστημα. Άρα λοιπόν, αν οι ποσοστώσεις μπορούν να χρησιμεύσουν για να αλλάξει το σύστημα, να τις χρησιμοποιήσουμε. Και πριν από λίγο η κυρία Πιατικάνεν έλεγε ότι έχει μείνει άναυδη, ότι μένει άναυδη όταν ακούει ότι κάποιοι θέτουν σε αντιπαράθεση τις ποσοστώσεις με την αξία. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε τις ποσοστώσεις για να προωθήσουμε ανίκανους ανθρώπους. Και γιατί θυμήσαμε και σήμερα το πρωί, μόνο για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ότι το 60% των πτυχιούχων πανεπιστημίου είναι γυναίκες. Προφανές λοιπόν είναι ότι δεν πρόκειται για ε, θέμα, δεν τίθεται θέμα αξιοκρατίας. Θέλουμε πραγματικά λοιπόν να ευχαριστήσουμε και εσένα για όλους τους αγώνες που έχει κάνει η Κομισιόν για τα δικαιώματα των γυναικών και για τα δικαιώματα γενικότερα των Ευρωπαίων πολιτών. σε καλωσορίζω και εγώ θερμά και έχεις το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους και σας χαιρετίζω όλους. Ξέρω πως έχετε δουλέψει πολύ εντατικά αυτές τις μέρες και πραγματικά βασιζόμαστε στη στήριξή σας, ε, στη στήριξη των εθνικών, μέσα στα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί η ισότητα των φύλων και η ισότητα γενικότερα στις κοινωνίες μας δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να ολοκληρωθεί και σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Και η Αντιπρόεδρος Αντζελίλη έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει εμεί να δώσουμε το σωστό παράδειγμα. Θυμάμαι ακόμη όταν ο πρόεδρος Βαρόζο έφτιαχνε την επιτροπή του, έπρεπε να συμφωνήσει με τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε τουλάχιστον να του υποβάλουν υποψηφίους έναν άντρα και μια γυναίκα, ώστε να έχει την επιλογή τουλάχιστον τα κατάφερε, ακόμα και αν όλες οι κυβερνήσεις δεν το έκαναν αυτό που του ζήτησε, κατάφερε να έχει 33% γυναίκες στην Επιτροπή. Δεν είναι το τέλειο, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας, να τακτοποιήσουμε το του οίκου μας, δηλαδή στη διοίκηση, στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαστε αυτή τη στιγμή στο 27 μόλις 100 γυναίκες και επειδή έχουμε ήδη ξεπεράσει το... Μάλλον δεν έχουμε μπορέσει να ξεπεράσουμε και να φτάσουμε το στόχο μας, θα τους αυξήσουμε ακόμη περισσότερο. Να σας πω δηλαδή ότι στη δική μου διοίκηση έχω 80% γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση και 60% στην μεσαία, στις μεσαίες θέσεις. Και καταλήγω στο ότι πραγματικά χρειάζομαι ποσοστώσεις, <laughs> ποσοστώσεις για τους άνδρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το γενικότερο θέμα μας σήμερα να έρθω αμέσω σε αυτά που θα θέλατε να συζητήσουμε, διότι έχουμε πραγματικό πρόβλημα στις κοινωνίες μας. Εντάξει, η δική μου γενική διεύθυνση δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση και όλοι το ξέρουμε. Το ξέρουμε από την εμπειρία μας στις χώρες μας και από την ευρωπαϊκή ε, εμπειρία το γεγονός ότι η Κομισιόν εργάζεται για ένα νομικό μέσο για την ισορροπημένη εκπροσώπηση για ανδρών γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών δεν προέκυψε εκ του μηδενό. Ξέρετε ότι γενικά προσπαθούμε να νομοθετήσουμε, μάλλον νομοθετούμε για την ισότητα των φύλων από τότε που φτιάχτηκε η Ευρώπη, γιατί αυτό είναι γεγραμμένο στις πρώτες συνθήκες, στις πρώτες συνθήκες του 57 της Ρώμης. Εκεί ήδη προβλέπονταν διατάξεις που απαγόρευαν τις διακρίσεις επί τη βάση του φύλου. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για όσους θέλουν να γνωρίζουν την ιστορία το πώς έγινε αυτό. Το 57 όταν ε, εκπονήθηκε η συνθήκη της Ρώμης, η πρόταση αυτή προέκυψε βασικά λόγω οικονομικών προβληματισμών. Η Γαλλία τότε ήθελε να εξαλείψει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστημένα στα διάφορα κράτη-μέλη. Και επειδή η Γαλλία ήδη είχε υιοθετήσει διατάξεις για ίση πληρωμή, ίσες αμοιβέ για άνδρες και γυναίκες, πολύ νωρίτερα από ό,τι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, φοβήθηκε ότι η φθηνή απασχόληση γυναικών, κυρίως στη Γερμανία, θα οδηγούσε τις εταιρείες να μετεγκατασταθούν και θα έθετε δηλαδή τις γαλλικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση. Αν δει λοιπόν κανείς την ιστορία βλέπει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Και μπορεί επίσης να θυμάστε ότι το 1979 το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε για το τότε άρθρο 119 της συνθήκης ότι ο στόχος δεν ήταν μόνο οικονομικός αλλά και κοινωνικός. Μέχρι το 1976, πριν δηλαδή να προσθέσει, προσθέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στις οικονομικές, στα οικονομικά συμφέροντα και τα κοινωνικά συμφέροντα, την κοινωνική πρόοδο και τη ε, βελτίωση των ε, συνθηκών διαβίωσης. Και ακόμα και σήμερα ο κοινωνικός και οικονομικός στόχος της ισότητας των φύλων είναι οι δύο, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Μπορεί να θυμάστε επίσης ε, την πολύ σημαντική απόφαση του δικαστηρίου του Μαΐου 1971 που αποτέλεσε την αρχή των όσων κάναμε τις επόμενες δεκαετίες. Ήταν η πρώτη απόφαση σε μια σειρά υποθέσεων που είχε διώξει η Γκαμπριέλ Ντεφρέν κατά του εργοδότη της της Σαμπένα ήταν πεύθυνη πτήση και διαμαρτυρήθηκε για άνεση αμοιβή στη εργασία. Και τότε διευκρινίστηκε ο στόχος της, νομοθεσίας, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί των φύλων και έλεγε ότι η αρχή της ίσης αμοιβή για ίδια εργασία είναι άμεσα εφαρμοστέα και πρέπει να ε, εφαρμοστεί και από τα εθνικά δικαστήρια. Αυτή ήταν η αρχή για τη σύγχρονη ισότητα των φίλων εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζετε μετά τη δεκαετία του 70 όλη την νομοθεσία που ακολούθησε για την ισότητα των φίλων στην απασχόληση, τις ίσες αμοιβέ, τις ε, προαγωγές, την κατάρτιση. Το επόμενο βήμα ήταν οι οδηγίες για την κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια και για τους ε, ανεξάρτητους επαγγελματίες, θα θυμάστε τους κανόνες για την αδιαμητρότητα, στη γονική άδεια και ούτω καθεξής. Αυτά για να σας πω ότι δεν, ε, δεν, δεν είναι κάτι το καινούργιο όλα αυτά. Είμαστε στη συνέχεια, στην ίδια πορεία για των όσων έχουν γίνει από γενναίες επιγενεών ανδρών και γυναικών στην ευρωπαϊκή πολιτική, από πολιτικούς και από δικαστές. Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι εκατοντάδες αποφάσεων που αφορούν την ισότητα αποτελούν μια νομολογία που έχει τεράστια σημασία. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα σε αυτή τη μακρά παράδοση. Η πρότασή μου λοιπόν για υποβολή ενός νομικού εργαλείου όσον αφορά την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών προσπαθεί να εγγυηθεί ότι η ισότητα ε, μεταχείρισης θα οδηγεί και στην πράξη σε ισότητα των φύλων και στην ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ιδέα των, των, των θετικών δράσεων που όλοι ξέρετε τι είναι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ισχύει στα κράτη-μέλη. Και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εδώ και δεκαετίες πια. Και τώρα συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 157 της Συνθήκης και αυτό που είναι νέο είναι ότι στο άρθρο 23 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε δηλαδή τη συνθήκη και όπως την είχαμε και πριν έχουμε το χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που ισχύει σαν Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έχουμε και πιο σημαντικό και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λέει λοιπόν ότι αυτές οι θετικές δράσεις θα έχουν στόχο να διορθώσουν την υφιστάμενη κατάσταση ανισορροπίας ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες σε συγκεκριμένους τομείς. Και όπως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυτές οι δράσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες και αναλογικές. Ας έρθουμε τώρα στο μέσο το οποίο προτίθεμε να προτείνω. Γιατί χρειάζεται επιτάχυνση η πρόοδος προς μια πιο ισόρροπη προσώπηση ανδρών και γυναικών στα πιο ψηλά αξιώματα. Διότι Γιατί είναι θέμα ισότητας βέβαια. είναι τα δικαιώματα και η οικονομία. Δεν είναι μόνο τα δικαιώματα. Αν το δείτε από οικονομικής απόψεως, είναι και πολύ συμφέρον το να υπάρχει ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Μια νομική δράση από πλευράς Ένωσης θα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και θα τονώσει και την απασχόληση και ε, την ανάπτυξη. Πού βασίζουμε όμως αυτή μας την ε, παραδοχή. Έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε πολλές μελέτες. Μια ολόκληρη σειρά και έπονται και άλλες. Και δεν είναι μη κυβερνητικών οργανώσεων ή πανεπιστημίων. Είναι μελέτες που κάνει ο ίδιος επιχειρηματικός κόσμος. Η Μακένζι, Ernest Young, Credit Suisse, ε, Deutsche Bank. Δεν είναι και περιβολικά φεμινιστικές αυτές οι οργανώσεις και οι τράπεζες και οργανισμοί. Και καταλήγουν όλοι στο ίδιο συμπέρασμα. Όσο περισσότερες γυναίκες έχουν οι εταιρείε στα διοικητικά συμβούλια, τόσο καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα έχουν. Με άλλα λόγια, όταν στις εταιρείε, στις μεγάλες ηγετικέ θέσει είναι γυναίκες οι εταιρείε αυτές παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και έχουν καλύτερη απόδοση και επιδόσεις και οικονομικά σε σχέση με άλλες που δεν έχουν. Γι' αυτό το λόγο, και γι' αυτό το λόγο μάλλον, η πρόταση ε, την οποία σήμερα επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποβληθεί μόνο από τον αρμόδιο επίτροπο για θέματα ισότητας των φύλων που είναι υποφαινομένη αλλά σε συμφωνία με τους ε, οικονομικούς επιτρόπους, τον κύριο Ταγιάννη, αντιπρόεδρο που είναι για θέματα βιομηχανίας, τον αντιπρόεδρο Ρεν που είναι για τα οικονομικά, τον επίτροπο Μπαρνιέ που ε, είναι επιφορτισμένος ε, ε, με τις εταιρείες και την εσωτερική αγορά και με τον επίτροπο Άντορ που είναι επίτροπος απασχόλησης. Βλέπετε, ένα προς τέσσερα, μία γυναίκα, τέσσερις άντρες. Λοιπόν, δικαιώματα ε, ισότητα και οικονομικά αποτελέσματα. Τα στοιχεία τα γνωρίζετε, τα δικά σας, στα κράτη σας. Σε ευρωπαϊκά επίπεδα τώρα, κατά μέσο όρο, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, έχουμε 86,5% άνδρες. Άρα το υπόλοιπο γυναίκες 13,5%. 97,5% των προέδρων είναι γυναίκες, μόνο 2,5% είναι άνδρες, συγγνώμη, γυναίκες, 2,5%. Ο μέσος όρος είναι αυτός, έτσι. Ε, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Ταυτόχρονα, ε, ακριβώ επειδή είναι τόσο λίγες οι γυναίκες, Είπαμε ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κατά 60% γυναίκες. Δηλαδή, Έχουμε ταλέντο, προσόντα, δεξιότητες, αλλά κάποια στιγμή αυτά δεν μεταφράζονται στην πράξη και δεν ακολουθούν ε, τους οικονομικούς ε, κύκλους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Ε, η ίδια η οικονομία έχει κάνει τις επιχειρήσεις, έχει κάνει τις μελέτες και οι εμπορικές σχολές, οι πιο σημαντικές ε, σε όλη την Ευρώπη, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν ένα κατάλογο γυναικών υψηλών προσόντων ε, με τα εφόδια που χρειάζονται και είναι έτοιμες να μπουν σε διοικητικά συμβούλια. Και έχουν και την εμπειρία και μπορούν από σήμερα να μπουν ε, στα διοικητικά συμβούλια. Μόνο 8.000 είναι αυτές οι γυναίκες. Ε, τα λαντούχες με υψηλά προσόντα υπάρχουν, είναι παρούσες, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να φτάσουν σε αυτά τα υψηλά αξιώματα, να ανέλθουν αυτή την κλίμακα. Και εμείς ως οικονομία έχουμε την ευκαιρία να εσωματώσουμε όλο αυτό το δυναμικό ε, στην οικονομία μας για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που αποδεικνύεται από τις μελέτες. Μόνο αν συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες, όχι μόνο στα πιο ψηλά επίπεδα, αλλά γενικά στην αγορά εργασίες, θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να αυξηθεί η απασχόληση ενηλίκων στο 75%. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν και οι γυναίκε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και τα δύο. Να εισέρχονται περισσότερες γυναίκε στην αγορά εργασία, αλλά και να καταλαμβάνουν τα ανώτατα αξιώματα. Για να λειτουργούν και ως πρότυπα, αλλά να έχουν και την ευκαιρία ανέλυξη ε, στα διαδρομία τους. Έρχομαι τώρα ε, το Μάρτιο του 2011 που προσκάλεσα τις εταιρείες να δεσμευθούν ε, εθελοντικά ε, με μια συμφωνία ε, εθελοντική να συμμετέχουν οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και ο στόχος είναι 30% μέχρι το 2015 και 40% μέχρι το 2020. Τι συνέβη έκτοτε. Σας είπα το 2011 έγιναν αυτά. Το 2012, ένα χρόνο ακριβώς μετά, κάναμε μια ανάλυση και ήρθε και την παρουσίασα και στο Κοινοβούλιο. Ήταν η ανάλυση της 5ης Μαρτίου του 2012, όπου θελήσαμε να μελετήσουμε αν αυτή η δέσμευση είχε υλοποιηθεί. Η υπόσχεση αυτή που ανέλαβε ο επιχειρηματικός κόσμος και αν υπήρχαν διαφορές ε, στις στατιστικές μας δώσαμε την ευκαιρία στην αυτορύθμιση, στην ε, εθελούσια επαναλαμβάνω. Αποτέλεσμα, υπήρξε μια αλλαγή, οφείλω να ομολογήσω, ε, διότι το 2011 ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών αυξήθηκε κατά 1,9%. Γιατί λέγω την αλλαγή αυτό, διότι τα προηγούμενα έτη είχε αυξηθεί μόνο κατά μισό της εκατό, μισή ποσοστία μόνο. Δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι είχαμε θέσει το θέμα επιτάπητος και είχαμε επίσης επιχειρήσεις, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε την αδράνειά σας. Κάντε κάτι. Βοήθησε αυτό για να ε, υπάρξει πιο γρήγορη εξέλιξη ή τουλάχιστον λιγότερο αργή σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, τι διαπιστώσαμε. Αυτή η αλλαγή, δηλαδή από το μισό της 100 στο 1,9% οφείλεται κυρίως στα κράτη-μέλη εκείνα που έχουν ποσοστώσεις στην νομοθεσία τους. 11 τον αριθμό. Στην Νορβηγία επιλέξαν πολύ διαφορετικές ε, λύσεις με νομική μορφή, μεταξύ αυτών και υποχρεωτικές ποσοστώσεις για να ενισχυθεί η γυναικεία παρουσία στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Είμαι βεβαία ότι εδώ έχουμε προσώπους από το Βέλγιο, τη Γαλλία ή την Ιταλία που εργάστηκαν στα κοινοβούλια τους για να εγκριθεί υποχρεωτική ποσόστοση. Άμεση λοιπόν συνέπεια αυτού του νόμου ήταν ε, τεράστια αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Και επίσης, οι άλλες χώρες, για να το πω ομά και ακατέργαστα, δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα σε αυτές τις χώρες, δεν έχει γίνει περίπου τίποτα. Στις ε, χώρες που δεν ανέλαβαν δράση έχει μείνει στάσιμη ή ακόμα και μειώθηκε η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και με την ταχύτητα αυτή θα χρειαστούμε δεκαετίες για να φτάσουμε μια σχετική ισορροπία και γι' αυτό όπως είπα πρέπει να δράσουμε τώρα. Η νέα πρόταση λοιπόν η οποία επίκειται θα οδηγήσει την Ευρώπη ένα βήμα περισσότερο στην προσπάθειά της να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να καταλήξει σε ένα ισόπεδο γήπεδο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα στην εσωτερική αγορά. Όσο εμείς συντάσαμε την πρόταση αυτή, ήμασταν υποχρεωμένοι να βασιζόμαστε και στις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Μία από αυτές τις αρχές είναι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα. Και ξέρω ότι και αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στη δική σας καρδιά ως εθνικών κοινοβουλευτικών. Έχουν ληφθεί υπόψη λοιπόν αυτές οι βασικές έννοιες. Θα σας δώσω έξι παραδείγματα για το πώς ελήφθη υπόψη. Ελήφθησαν υπόψη δύο αυτές αρχές. Ένα. Η πρόταση αφορά μονάχα την, ε, το ποσοστό των γυναικών που είναι στα διοικητικά συμβούλια αλλά δεν έχουν εκτελεστικές λειτουργίες στις εταιρείες τους. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην εσωτερική διαχείριση και στις εσωτερικές διαχειριστικές αποφάσεις των εταιριών, γιατί αυτό μπορεί να αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεύτερον, το νομικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να αφορά μόνο εταιρείε που είναι εισηγμένε στα χρηματιστήρια εκτός από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και αν εισηγμένε στα χρηματιστήρια. Τρίτον, θα πρέπει τα, τα προσόντα να είναι το αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Αν λοιπόν είναι θέμα προσόντων θα πρέπει να διαλέγουμε γυναίκες λόγω των προσόντων της και όχι λόγω του φίλου της. Δεν θα πρέπει ποτέ να βάζουμε μια γυναίκα σε μια θέση ηγετική μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό επειδή είναι καλές, επειδή έχουν τα προσόντα. Το κείμενο λοιπόν αυτό προβλέπει ότι το φύλλο το οποίο υποεκπροσωπείται θα πρέπει να έχει μια ευκαιρία να προωθηθεί περισσότερο για να επιτευχθεί η ισορροπία. Επίσης έχουμε και μια ρήτρα ευελιξίας Αν σε μια επιχείρηση δεν είναι δυνατό από την οπτική γωνία του εργοδότη να βρει ένα υποψήφιο από το φύλλο που υποεκπροσωπείται, διότι δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφοι, τότε υπάρχει δυνατότητα ευκαμψίας, να εφαρμοστεί μια ρήτρα ευκαμψίας. Πέμπτο στοιχείο οποιαδήποτε νομοθεσία περί ποσοστώσεων θα πρέπει να είναι μεταβατικού χαρακτήρα, προσωρινή. Υπάρχει μια ρήτρα εκπνοής, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να έχουμε στο δινεκές μια ποσόστοση. Απλώς να σπάσουμε τη γυάλινη οροφή που αναφέραμε προηγουμένως. Και άμα τη σπάσουμε και την κάνουμε ρημαδιό, δεν χρειαζόμαστε πια ποσοστώσεις. Είναι ένα προσωρινό λοιπόν μέτρο για να περάσουμε, να ξεπεράσουμε αυτό το φραγμό. Και το έκτο σημείο σε σχέση με τις κυρώσεις, τα κράτη-μέλη θα πρέπει από μόνα τους να επιλέξουν από μία σειρά κυρώσεων που ισχύουν ήδη στην Εθνική Νομοθεσία σε ορισμένα κράτη-μέλη, με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουν κυρώσεις σε εταιρείε οι οποίες δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία αυτή για την επίτευξη της ισότητας. Πιστεύω λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για σας που είστε μέλη των αρμοδίων επιτροπών ισότητα στα Εθνικά Κοινοβούλια να γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία της πρόταση της Κομισιόν, γιατί τα στοιχεία αυτά θα τύχουν συζήτηση από τους συναδέλφους σας στη Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σας ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Κοινοβουλίου σας όταν αναλύουν τα θέματα επικουρικότητος για την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτό είναι φιλική προς την αρχή της επικορικότητα αυτή η πρόταση. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει εσείς να επισημάνετε στο δικό σα κοινοβούλιο ως γνώστριες αυτής της νομοθεσίας. Και επειδή η επικορικότητα παραμένει μια γενική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου, γενική αρχή που σημαίνει ότι πρέπει πάντα τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται στο λιγότερο κεντροποιημένο επίπεδο νομοθεσίας που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τη δυνατότητα να νομοθεστήσουμε μόνο αν σε εθνικό επίπεδο ή σε υποδέστρο επίπεδο δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Και κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετεί στον τομέα της ισότητας των φύλων ή στον τομέα του εταιρικού δικαίου, όπου και εκεί υπάρχει μια μακρά ιστορία από το 1969 νομοθετημάτων, παραδείγματος χάρη η εταιρική ε, διακυβέρνηση για λογιστικά πρότυπα κτλ. Η πρότασή μας λοιπόν θα πράξει το ίδιο, θα άπτεται του εταιρικού δικαίου και θα ενισχύσει αυτά τα οποία υπάρχουν ή είναι υπό εξέταση σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά σε εθνικό επίπεδο μπορεί κανείς να υπερκεράσει αυτά τα οποία προτείνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου και προς όφελος της εσωτερικής αγοράς, το νομοθέτημα αυτό θα δημιουργήσει ένα ε, ίσο πεδίο ανταγωνισμού για όλες τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείε, γιατί αυτές είναι κυρίως οι εταιρείε οι οποίες εμπλέκονται σε διαμεθοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες. Η πρόταση είναι ακόμα υπό εξέταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων. Όλα αυτά τα οποία σας είπα είναι κατά πόσο πιθανότητα το πιθανό περιεχόμενο αυτής της πρότασης, αλλά όταν περατωθεί αυτή η πρόταση θα είμαι έτοιμη να έρθω ενώπιόν σας και να συζητήσω μαζί σας για το περιεχόμενο αυτής της πρότασης και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βασιστώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόλυτα και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι μπορώ να βασιστώ και στα Εθνικά Κοινοβούλια για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό και να μπορέσουμε να το φέρουμε σε αίσιο πέρας γιατί είναι απαραίτητη αυτή η νομοθεσία για την κοινωνία μας και είναι απαραίτητη και για την οικονομία μας. Θα προσπαθήσω να μιλήσω ειδικά εγώ τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε, κύριε Ρέντινγκ. Με πολύ μεγάλη σαφήνεια σκιαγραφίσατε το ιστορικό πλαίσιο και υπόβαθρο αυτής της υπόθεσης. Και είναι επίσης ε, σημαντικό να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα για να κατανοήσουμε ε, και την όλη υπόθεση. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη αφοσίωσή σας και φαίνεται καθαρά ότι το θέμα σας ενδιαφέρει και προσωπικά. Ξέρω ότι πρέπει να αποχωρήσετε αρκετά γρήγορα. Να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Ο κύριος Ρωμέβα, πολύ σύντομα στα αγγλικά. Ε, σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας. Γνωρίζετε ότι στο Κοινοβούλιο έχετε πολύ καλούς όσο και ισχυρούς συμμάχους και θα ε, δώσουμε αυτή τη μάχη όπως ζητήσατε. Κάτι που συνδέεται όμως με τις ίσες ευκαιρίες. Η αυτό που ονομάζουμε ισομερή εκπροσώπηση. Παράλληλα γίνεται μια συζήτηση για τη μείωση της μισθολογικής ψαλίδας. Ξέρω ότι το συζητάτε και αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας. Το Κοινοβούλιο εγκρίναμε ένα ψηφισμά πριν από μερικούς μήνες, ειδικά για αυτό το θέμα, για την αναδιατύπωση της οδηγίας, για την ίση αμοιβή και ανησυχούμε, ξέρετε, λίγο, γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπουμε να κινούνται τα πράγματα, ούτε λαμβάνεται υπόψη τόσο γρήγορα όσο ζητούσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του εκείνο. Θα μπορούσατε λίγο να μας διαφωτίσετε σχετικά. Ε, we take one more... Ε, Άλλη μια ερώτηση και μετά να απαντήσει. Βουλευτές και ευρωβουλευτές, ένα To Mrs. from Germany. Η κυρία Λάουριχ από τη Γερμανία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με μεγάλο ενθουσιασμό σας ακούω εδώ, κύρια Ρέντινγκ, γιατί και στη Γερμανική Βουλή και στην Επιτροπή μας είπατε τα ίδια. Είστε πάρα πολύ αποφασισμένοι να προωθήσετε αυτή την υπόθεση της συμμετοχής των γυναικών και αναγνωρίζεται και μια μεγάλη ανάγκη ε, στην πολιτική ισότητα. Ε, αυτό που μας είπατε σημειώνω, θα τα διαβιβάσω στην Επιτροπή μου, αλλά δεν σας κρύβω ότι η συζήτηση στη Γερμανία είναι πάρα πολύ επίμαχη. Γι' αυτό πιστεύω ε, χρειαζόμαστε σαφή μηνύματα από τις Βρυξέλλες, αλλά και από το σύνολο της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η δυνατότητα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής στο μέλλον θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί η πολιτική ισότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τις ποσοστώσεις, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ κεντρικό, ε, αφιερωνόμαστε σε αυτό και θα έρθουμε εδώ με την Επιτροπή μας ε, να σας επισκεφτούμε την άλλη εβδομάδα και σίγουρα θα ε, πρέπει να προωθήσουμε μία στεναρή και αποφασιστική πολιτική ισότητας ε, στα κράτη-μέλη, στα διάφορα κοινοβούλια και να τα διαβιβάσουμε. Αυτά προς το παρόν ως δήλωση και σας ευχαριστώ. President, uh, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Να αρχίσω με τη δική σας ερώτηση, κυρία Λάουρισκ. Ξέρω πως είναι πολύ επίμαχο αυτό το θέμα, αλλά είναι και ζήτημα πολιτικής ηγεσία. Αν οι πολιτικοί κάνουμε μόνο ό,τι δεν είναι αντιφατικό και επίμαχο, α, τότε ας πάμε σπίτια μας. Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που είναι απαραίτητο και, και σημαντικό. Εδώ και χρόνια προσπαθούμε και ξέρουμε πως δυστυχώς δεν γίνεται χωρίς νομοθεσία. Και γι' αυτό λέω πως δεν θεωρώ αυτή τη νομοθεσία ως στόχο, αλλά ως ένα μέσο για να σπάσουμε το κρυστάλλινο, την κρυστάλλινη αυτή οροφή θα βάλουμε μια προθεσμία, μια, μια ημερομηνία όπου αυτή η νομοθεσία αυτό, αυτόματα θα ε, καταργηθεί και θα έχει μεγάλο αντίκτυπο πολύ σύντομα γιατί το γυναικείο ταλέντο υπάρχει, είναι διαθέσιμο πολύ γρήγορα. Αυτό το ίδιο το γυναικείο ταλέντο θα θα αρχίσει να λειτουργεί. Και σε σχέση με το μισθολογικό, τη μισθολογική ψαλίδα έχουμε οδηγία από το 2006. Και αυτή τη στιγμή αναλύω πώς εφαρμόστηκε αυτή η οδηγία και επιβλήθηκε στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα επανέλθω με έκθεση για αυτό το θέμα πολύ σύντομα, το 2013, μέσα στο 2013, και επί τη βάση αυτής της έκθεσης, όταν θα δούμε πια πολύ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα πού έχει μειωθεί πρόοδος και πού όχι, τότε θα μπορέσουμε ίσως να τη διορθώσουμε, να φτιάξουμε καινούργια ε, νομοθεσία, καινούργια οδηγία. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Συνεχίζουμε με την αύξηση της ενημέρωσης, ε, και δραστηριότητες για την ίσες αμοιβέ και για την μισθολογική ψαλίδα, για την κατάρτιση και την προετοιμασία εργαλειών για τις εταιρείε, ε, κατάρτιση για εκείνα τα μέλη των εταιριών που ενδιαφέρονται για αυτού του είδος τις πολιτικές. Ξέρετε επίσης πως η Κομισιόν έχει φτιάξει και μια Ευρωπαϊκή ημέρα ίσης αμοιβή. Φέτος ήταν στις 5 Μαρτίου. Και γιατί στις 5 Μαρτίου? Γιατί μέχρι τις 5 Μαρτίου οι γυναίκες έπρεπε να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται. Λόγω της μισθολογική διαφοράς. Και πληρώνονται μόνο από τις 5 Μαρτίου και έπειτα. Βεβαίως κατά μέσο όρο είναι αυτά τα νούμερα, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό να δούμε πόσο περισσότερο μια γυναίκα πρέπει να δουλέψει πριν να φτάσει στο επίπεδο των μισθών. 62 μέρες για την ώρα είναι η διαφορά. Μια φορά ετησίως επίσης διοργανώνουμε και ένα φόρουμ για να ανταλλάξουμε γνώσεις με όσους εργαζόμενους και συνδικαλιστές εργάζονται στον τομέα όπου υπάρχουν οι πληροφορίες δεν είναι κάτι το οποίο αφήνουμε, το δουλεύουμε διαρκώς. Αλλά η ανάλυση των όσων έχουν γίνει θα είναι εδώ ε, επιτάπητος σε αυτό το σώμα το χρόνο. Κυρία Κοχμαρίνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ κυρία Ρέτιν για την παρουσία σας και για το θάρρος το οποίο έχετε δείξει στο πολιτικό για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην πρότασή σας. Βλέπουμε βέβαια ότι πολλοί από εμά ε, είμαστε ενοχλημένοι από το γεγονός ότι δεν έχουν ευδοκιμήσει τα εθολοντικά μέτρα. Και εξάλλου η πρότασή σας αφορά τα διοικητικά συμβούλια αλλά όχι το εκτελεστικό τμήμα των εταιριών. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρότασή σας, κατά την άποψή μου, είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Έχει υπάρξει μια συζήτηση τόσο μακρά που ορισμένοι έχουν ξεχάσει την ε, αρχή αυτής της συζήτησης. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο έχει γίνει χωρίς καμία ε, προετοιμασία. Υπήρξαν πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Ευρώπη, πάντα με τις ίδιες ε, προθέσεις, τις ίδιες δηλώσεις ότι τα οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν το έργο να προχωρήσουν στον τομέα αυτό, αυτό τελικά δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι πραγματικότητα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και κίνηση σε νομοθετικό επίπεδο και όπως είπε η κυρία Λάτσεκ από την γερμανική Bundestag το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενο στη Γερμανία αλλά αυτό καταδεικνύει και πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πόσο είναι απαραίτητο να κινηθούμε με ένα συνεπή και συνεκτικό τρόπο. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς έχουμε υποστηρίξει πολλές φορές και με υποστηρίξει 80% των βουλευτών έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις στον τομέα αυτό. 80% λοιπόν των βουλευτών έχουν πει στην Κομισιόν ότι περιμένουμε να έχετε μια νομοθετική πρωτοβουλία για την επίτευξη ισότητας στον τομέα αυτό και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορεί το θέμα αυτό να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η φιλελεύθερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάντα υποστηρίξει αυτέ τι ενέργειε και θα συνεχίσει να τι υποστηρίζει. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, η γερμανική Bundestag, ή μάλλον η νομική υπηρεσία της ε, Bundestag έχει πει ότι είναι σύμμορφη μια τέτοια πρόταση με το γερμανικό βασικό νόμο και δεν πρόκειται να αντιταχθεί σε κάτι τέτοιο. Εμείς τώρα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ενοχληθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιδράσει το Συμβούλιο και πώς μερικά κράτη-μέλη βολεύονται να ξεχνούν τι λέει η συνθήκη σε σχέση με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Εμείς ε, περιμένουμε την ε, ε, περιμένουμε την επίσημη πρόταση, δεν θέλουμε όμως να, το Συμβούλιο την απορρίψει προτού καν δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας υπενθυμίσατε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπήρξε πραγματικά μια μακρά προπαρασκευαστική διαδικασία για αυτό το νομοθέτημα. Δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε μία αγορά ελαφρά την καρδία. Αν παρέμβει κανείς σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι αποχρόντες λόγοι και πρέπει ο στόχος της παρέμβαση αυτή να είναι προς το όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας Και αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Δεν μπορεί να κάνει κανεί λοιπόν χωρίς προετοιμασία μια τέτοια παρέμβαση. Αλλά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν, έχουν συλλεχθεί. Είναι φανερό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις σε ψηφίσματά του ζητήσει από την Κομισιόν να αναλάβει δράση. Η Κομισιόν λοιπόν επεξεργάζεται το κείμενο του νομοθετήματος και προβλέπω ότι το κείμενο αυτό θα σας δοθεί, εν... σας δοθεί σύντομα και μετά θα ακολουθηθεί η φυσιολογική διαδικασία στα θεσμικά μας όργανα, θα εξεταστεί από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και οι δύο συν νομοθέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν σε σχέση με το τελικό κείμενο το οποίο θα έχει τον χαρακτήρα νόμου. Θα θυμόσαστε πράγματι την παράξενη αυτή επιστολή κάποιων πρεσβευτών από τα κράτη-μέλη που θέλαν να εμποδίσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να, να την αποτρέψουν από το να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Εν τω μεταξύ υπήρξαν πολλές άλλες επιστολές και από άλλα κράτη-μέλη που λένε ότι είναι πολύ καλή πολιτική να ακολουθήσει η Κομισιόν αυτή που προτείνεται και σας αναφέρω μονάχα μία επιστολή για την ενδιαφέρουσα. Είναι η επιστολή της γαλλικής κυβέρνησης. Το περιεχόμενο είναι θετικό σε σχέση με την πρωτοβουλία της Κομισιόν. Αυτό το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον είναι η υπογραφή αυτού του γράμματος. Έχει δύο, φέρει δύο υπογραφές αυτή η επιστολή. Την υπογραφή του Υπουργού για Ισότητα Ευκαιριών, που είναι μια γυναίκα, και επίσης την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών Θεμάτων, που είναι άντρας. Πολιτικά λοιπόν αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει πράγματι αυτή η εξισορρόπηση μεταξύ των ίσων ευκαιριών από τη μία πλευρά και των υπευθύνων για τον οικονομικό αντίκτυπο από την άλλη πλευρά που πρέπει να εξισορροπηθούν αυτές οι δύο ε, πλευρές και να το πράξουμε με έναν τρόπο που να, είναι, να συνάδει με την ευρωπαϊκή πολιτική ότι όλοι αυτοί που πρέπει να είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να, είναι, εργαστούν από κοινού. Μπορεί να είναι γυναίκες, μπορεί να είναι άντρες και αυτή η συνεργασία αποδίδει τους καλύτερους καρπούς. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευτυχής που μαζί, και μαζί και με την κυρία Αντζελίλη που μπορέσατε να βρείτε χρόνο για να παρακολουθήσετε την διάσκεψή μας και να ήρθε εδώ μαζί μας. Ξέρω πως πρέπει να φύγετε, πως έχετε άλλες ε, υποχρεώσεις. Είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε. Και να ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σας. Då Και τώρα συνεχίζουμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Ασαλάνη από την, ε, από την Σουηδία. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς η κυρία Επίτροπος έφυγε, ήθελα να της θέσω ένα ερώτημα, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Αντζελίλη, την αντιπρόεδρο Αντζελίλη και τον πρόεδρο Γκούστευσον. Εμεί είχαμε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία που παρακολουθήσαμε στην Ορβηγία σε σχέση με τις ποσοστώσεις για τα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχουν ορισμένες γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε πολλά διοικητικά συμβούλια αυτό δεν είναι βέβαια μεγαλύτερη συμμετοχή ε, γυναικών. Πώς μπορούμε λοιπόν με την πρόταση της Κομισιόν να ξεπεράσουμε προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην παράκαμψη του συστήματος ε, ποσοστώσεων, γιατί και στη Σουηδία αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα και για μας ως βουλευτές του Σουηδικού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της πρότασης ε, της Κομισιόν και θα θέλαμε να ξέρουμε και ποια, ποιες είναι οι προθεσμίες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση για να μπορούν να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ηγεσία στην ε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούνται και με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια των ε, Ευρωπαίων φορολογουμένων για να εξασφαλίσουν αυτή την ισορροπία. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι η ενίσχυση των ε, ρυθμίσεων για την πρόληψη των ε, διακρίσεων, γιατί κοστίζει πολύ η δράση κατά των διακρίσεων. Μια άλλη πτυχή, η οποία δεν ακούστηκε σε αυτή τη συζήτηση, είναι οι προοπτικές για τις νέες γυναίκες. Τις νέες γυναίκες που έρχονται στην αγορά και που θα είναι οι αυριανές υπεύθυνε για τη λήψη αποφάσεων. Για την ώρα αυτοί που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή είναι μεσήλικες ή και ηλικιωμένοι. Το λέω με όλο το σεβασμό. Αλλά πρέπει να απασχοληθούν και νέοι. Νέοι άνδρες και γυναίκες, γιατί αυτοί θα αποφασίζουν για την πολιτική περισσότητα του μέλλοντος. Ναι, ε, και λυπάμαι γιατί όσοι θα πάρουν τώρα το λόγο δεν, θα έχουν, δεν, δεν μπορούν άμεσα να θέσουν τις ερωτήσεις στην κυρία Ρέντινγκ, ε, γιατί έφυγε και λυπούμε γι' αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε εμείς με τον κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Τόμσεν δεν είναι πια εδώ ό,τι φαίνεται. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι εδώ από τον κατάλογο που έχουμε φτιάξει. Η κυρία ε, Πέσκομετ από την Ολλανδία. Συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σας. Ευχαριστώ. Κρίμα που έφυγε η κυρία ε, Ρέντινγκ, πιστεύω κι εγώ, γιατί θεωρώ το θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό να ανταλλάσσουμε απόψεις από αυτών των ζητημάτων μιλάω αγγλικά και ακούω την Ολλανδική μετάφραση των όσων λέω. Λοιπόν, ε, συνεχίζω. Ήθελα να κάνω ερωτήσει στην κυρία Ρέντινγκ. Εμείς υποστηρίζουμε στην Ολλανδία αυτή την προσπάθεια για τις ε, γυναίκες στα Δυτικά Συμβούλια και ε, το 2009 σχεδόν ομόφωνα περάσαμε μια εθνική νομοθεσία για να είναι 30% στα διοικητικά συμβούλια αλλά και στα εποπτικά συμβούλια των επιχειρήσεων γυναίκες. Η εθνική μας νομοθεσία βασίζεται στην αρχή εφαρμόζηση εξηγής, comply or explain. Από την 1η ε, του 2016 ε, θα σταματήσει. Είναι, είναι προσωρινή δηλαδή αυτή η λύση. Και κινούμε από την παραδοχή ότι είναι ένα θέμα ευθύνη των κρατών μελών αυτό. Οι εθνικέ εταιρείε ε, πρέπει να ασχολούνται με αυτό, οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι. Και η πλειοψηφία τη Βουλή μα ε, είναι κατά των ευρωπαϊκών δεσμευτικών ποσοστώσεων. Μπορεί να ακούγεται ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, οπότε ας αλλάξουμε το σύστημα. Αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Εγώ είμαι φιλελεύθερη πολιτικός και εγώ, όπως η προλαλήσασα, και η ιστορία μας έχει διδάξει ότι το να αλλάξει κανείς νοοτροπία δεν γίνεται με αλλαγή συστήματος. Η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας γίνεται από τους ανθρώπους τους ίδιους. Και θα πρέπει να η πίεση να έρχεται από κατά κάτω, όχι από πάνω. Μόνο τότε έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις το παιχνίδι. Αυτά ήθελα να σας πω εξ ονόματος της Ολλανδικής Βουλής και ελπίζω η κυρία Ρέντινγκ να ενημερωθεί για αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ξανά ότι το θεωρώ μεγάλο κρίμα και εγώ εξεπλάγει που έπρεπε να φύγει πριν τις 4.30 η κυρία Ρέντινγκ. Δεν το ήξερα προηγουμένως. Κανονικά έπρεπε να παραμείνει. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Έφυγε η γυναίκα. Δεν μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις. Λυπάμαι και εγώ πάρα πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο, εξ όσων ε, βλέπω εδώ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι... κανονικά μπορούμε να τελειώσουμε δύο λεπτά νωρίτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Ωραία. Και έρχομαι τώρα στο συμπέρασμα της συνεδρίασης. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Αντιπρόεδρο ε, για να κλείσει. Αλλά προηγουμένως να πω μερικά πράγματα εγώ. Ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα σήμερα Εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα εξή και θα ήθελα να σας τα αναφέρω. Υπόθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να συμφιλιώνει τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο. Σωστό είναι αυτό και σημαντικό. Και πολλοί είπαν ότι εμείς εδώ ακριβώς στα θεσμικά όργανα θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Όταν μιλούμε για ισότητα και πόσο σημαντική είναι και πώς ε, συμφιλιώνεται η επαγγελματική ζωή με την ιδιωτική, θα πρέπει να αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο εσωτερικό τους να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τους ίδιους τους υπαλλήλους και να έχουν αυτή την ευκαιρία. Ε, τα όσα πρεσβεύουν δηλαδή τα θεσμικά όργανα τα εφαρμόζουν. Αλλιώς δεν γίνεται. Ε, ένα άλλο όπου ακούσαμε, η φροντίδα των παιδιών, η ειδική σταθμή κτλ. Και γιατί πάντα αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα που συνδέεται με τις γυναίκες. Συμφωνώ, είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, είναι στρεβλή η οπτική γωνία. Είναι ένα θέμα που αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες. Ε, ποιος θα φροντίζει τα παιδιά, αλλιώς δεν μπορεί να δουλεύει κανένας από τους δύο. συζητήσαμε και για τις διάφορες δομές, το είπα και προηγουμένως, ε, το πρωί. Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Όταν δουλεύει ένας γονέας, ο ένας από τους δύο είναι συνήθως ο άντρας. Και όταν υπάρχουν παιδιά προσχολικής ε, ηλικίας χωρίς φροντίδα, κάθεται η μαμά του στο σπίτι και δεν δουλεύει. Μα γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η φροντίδα των παιδιών για να μπορούν καν να εισέρχονται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Έτσι έχει η κοινωνία μας, έτσι είναι οι δομές οι κοινωνικές, όσο στρεβλή και λάθος. Είναι, είναι αυτό το πρότυπο στην κοινωνία, στην πολιτική ισότητα. Στη Σουηδία ένα από τα βασικά που κάναμε ήταν η προσχολική ε, ε, ηλικία και η παιδική και βρεφονιπιακή σταθμή. Ε, αφόσον αναπτύχθηκαν αυτοί, έγιναν οι γυναίκε ανεξάρτητες οικονομικά, βγήκαν στην αγορά εργασία και έχουν τελείως διαφορετική συμμετοχή στην κοινωνία. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντική η μεταρρύθμιση και για τις γυναίκες και για τους άνδρες, αλλά κυρίως για τι γυναίκε. Και επίσης πιστεύω πάρα πολύ στη γονική άδεια. Γονική είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς ε, πώς έχει η οικογενειακή ζωή χωρίς γονική άδεια. Είναι αρκετά άκαμπτη και αυστηρή η ε, ρόλη ε, των γονέων που εργάζονται και οι δύο. Ακόμα και όταν δεν δουλεύει η γυναίκα, η εργασία είναι και αυτή παρόλο που δεν αμείβεται. Και ε, θα πρέπει να μοιράζεται κανείς αυτή την εμπειρία. Εγώ το έχω ζήσει. Τη γονική άδεια την πήρα μισή-μισή με τη γυναίκα μου. Και πραγματικά έτσι έχουμε και καλύτερη εικόνα για το τι σημαίνει να είσαι σπίτι και να φροντίζεις τα παιδιά σου. Ε, ε, να δουλεύεις. Και ένα τελευταίο γιατί εκπροσωπούνται τόσο λίγο οι γυναίκες στην πολιτική. Και αυτό έχει να κάνει με τα πρότυπα και τους ρόλους. Ότι οι άνδρες ε, προτείνουν άνδρες υποψηφίους, ψηφίζουν άνδρες και εκλέγονται άνδρες. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, τελευταίο, ε, αυτή η εκστρατεία 50-50, που πρότεινε η κυρία Πιετικάινεν, πολύ σημαντική καμπάνια και μας επιτρέπει να είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και εν ώψη ενδεχομένω των ε, ευρωεκλογών να αρχίσουμε μια τέτοια εκστρατεία. Ελπίζω όλοι να, συμφέρετε, να συνεισφέρετε συγγνώμη, στη χώρα σας. Πολύ καλή αυτή η διάσκεψη. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Αντζελίλη για την πρωτοβουλία της διάσκεψης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους προσωπικά γιατί ήταν πάρα πολύ ε, καλή και θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό και τους υπαλλήλους, γιατί ξέρετε ότι τη δουλειά εδώ δεν την κάνουν οι βουλευτές, αλλά κάποιοι αφανείς ε, υπάλληλοι, ήρωες που αν δεν ε, εργαστούν δεν μπορούμε εμείς να συνεδριάζουμε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και εσάς τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, όλους ιδιαίτερους που ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας τις απόψεις σας. Θέλω να ευχαριστήσω και όλου του διερμηνεί, λέει ο Πρόεδρο. Έχει την καλοσύνη, γιατί χωρίς τους διερμηνεί δεν μπορούμε να συνεννοούμαστε καν. Ευχαριστώ πολύ. Grazie Presidente, io sono già intervenuta più di una volta. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πήρα το λόγο πολλές φορές. Θέλω απλά να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες, να υπογραμμίσω ότι ε, τούτο εδώ θα πρέπει να είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς, όχι μόνο διασκέψεων, αλλά επαφών, ανταλλαγών απόψεων, ε, γιατί πιστεύω πως αυτός είναι ένας ε, πολύ χρήσιμος και επικοδομητικός τρόπος για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, καλές πρακτικές και να συνεργαζόμαστε εν γέννη. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Και θα τρέξω κι εγώ τώρα, <laughs> γιατί όντω προσπαθώ να συνδυάσω την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή και σε λίγο πρέπει να πάρω το αεροπλάνο να πάω σπίτι μου. <laughs> Σας ευχαριστώ.